Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to open. Αγαπητοί. συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να κηρύξω την έναρξη της σημερινής συνεδριάσεως. Πρώτα απ' όλα, έγκριση της ημερήσια διάταξης. Συμφωνούμε με το σχέδιο ημερήσια διάταξης. Παρακαλώ, κύριε Φανίστερόη. Ευχαριστώ πολύ. Δύο πράγματα. Τι δευτέρε, όταν έχουμε ψηφοφορία, ίσω θα ήταν καλύτερα να τι βάζουμε λίγο αργότερα στην ημερήσια διάταξη και όχι στην αρχή-αρχή, γιατί μερικέ φορέ δεν προλαβαίνουν να έρθουν εδώ οι βουλευτέ και να είναι όλοι εδώ στι 3. Δεύτερον, πιο συγκεκριμένο, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τα δύο σημεία, 4 και 5 δηλαδή, γιατί κάποιοι συνάδελφοι μου ζήτησαν, μπορούμε να βάλουμε πρώτα το 5 και μετά το 4. Ευχαριστώ. Για την ψηφοφορία πρέπει να σας πω ότι προσπαθούμε να βάζουμε πάντα μια συγκεκριμένη ώρα που θα γίνει η ψηφοφορία, γιατί έτσι είναι πιο εύκολο για όλους. Αυτό είναι ο λόγος. Το 3 είναι συγκεκριμένο. Τώρα για την, ε, το άλλο που ζητήσατε, οι συγητές συμφωνούν, υπάρχει καμιά αντίρρηση. Παρακαλώ κύριε Φαν εγώ προτιμάω να κρατήσουμε την ημερήσια διάταξη ως έχει, γιατί σε μία ώρα περίπου πρέπει να φύγω, να ψηφίσουμε και μετά είναι το δικό μου θέμα να το αφήσουμε ως έχει, παρακαλώ. Πρόεδρος, καλώς. Συνεπώς θα ακολουθήσουμε την ημερήσια διάταξη ως έχει και δεν θα προβούμε σε αλλαγές. Καλώς. Αυτό θα κάνουμε. Τώρα δεν έχω ανακοινώσει τη Προέδρου. Έτσι κι αλλιώ τις κάναμε πριν από λιγότερο από μία εβδομάδα, δεν έγινε και τίποτα στο μεταξύ. Το μόνο που έγινε είναι ότι όλοι οι συγητέ και συντάκτες δούλεψαν πολύ σκληρά. Και περνάμε στην ψηφοφορία. Σήμερα έχουμε ψηφοφορία της γνωμοδότησής μας που είναι για τη θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα live. Συντάκτρια γνωμοδότησης για μας είναι η κυρία Μαρία Γκαμπριέλια Τζοάνα. Γνωρίζετε την ιστορία. Παρουσίασε το σχέδιο κειμένου της η κυρία Ζωάνα στις 13 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή μας. Ε, πρέπει να εξετάσουμε 98 τροπολογίες που υποβλήθηκαν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την εισηγήτρια και από ευρωβουλευτές και υπάρχουν 17 συμβιβαστικές τροπολογίες μετά από διαπραγματεύσεις. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ψηφίσει τη δικιά της έκθεση τον Νοέμβριο. Οπότε προλαβαίνουμε. Δεν βλέπω εδώ την κυρία Τζοάνα. Φτάνει, ε, φτάνει, είναι στο δρόμο. Στη Ρουμανία έχει μία διάσκεψη γι' αυτό, αλλά θα έρθει. Ωραία, έτσι ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα της κυρία Ζώνα. Η αλήθεια είναι ότι στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής μας ήταν ιδιαίτερα δραστήρια. Τότε πάρα πολλοί ευρωβουλευτές ήταν απόντες. Εκείνο όμως ήταν εκεί και τα εξήγησε όλα. Εκείνη ήταν εδώ. Λοιπόν, σήμερα ψηφίζουμε τη γνωμοδότησή της. Περνάμε στην ψηφοφορία.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 αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 82 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 83 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 87. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88. Με προφορική τροποποίηση. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροποποίησης? Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την 88 με την τροποποίηση. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 98 τώρα υπέρ, η 97 καταπίπτει, επειδή εγκρίθηκε 96. 98 λοιπόν τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ,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 εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία που θα γίνει ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα τη ψηφοφορία. Και η γνωμοδότηση εγκρίθηκε. Σε χαρητήρια και ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης. Στη συνεδρίασή μα στι 27 Σεπτεμβρίου είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την ε, θέσπιση ενός ε, μηχανισμού μέσα στον οποίο θα μπορούσαν ε, οι αρχές να συμφωνήσουν για την εφαρμογή και σε διασυνοριακά project. Ο μηχανισμός λοιπόν νομικών και διοικητικών διατάξεων ενός κράτους. Στόχος είναι να μειωθεί η διοικητική πολυπλοκότητα που καθυστερεί πολλές φορές πολύτιμα δυσυνοριακά project. Ο κύριος Φαν Μίλτεμπουργκ θα μας παρουσιάσει σήμερα το σχέδιο έκθεσής του. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία ανταλλαγή απόψεων. Η συζήτηση ήταν άκρος ενδιαφέρουσα. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πρόκειται για έναν από τους ε, τέσσερις νομοθετικούς φακέλους ε, για τους οποίους είναι αρμόδια επιτροπή μας. Κύριε Φαν Μίλτεμπουργκ, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω στο Λονδικά, λέει ο κύριος Μίτελμπεργκ. Αν μου επιτρέπετε, οπότε φορέστε τα ακουστικά σας. Πρόεδρε, όπως σωστά το είπατε, συζητάμε και πάλι, έχουμε και πάλι ανταλλαγή απόψεων για την δυνατότητα που υπάρχει διασυνοριακού μηχανισμού μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν ακριβώς ε, μηχανισμό σε διασυνοριακό πλαίσιο. Πρόκειται δηλαδή για πρόθεση της συνεργασίας, της διασυνοριακής συνεργασίας με έναν μηχανισμό ο οποίος μπορεί να βοηθήσει να καταλήξουν σε λύσεις διασυνοριακές περιφέρειες εφόσον αντιμετωπίζουν εμπόδια εξαιτία αυτής της παραμεθόριας διάστασης για να φέρουν σε πέρας κάποιο έργο. Σε αυτό πρέπει να συμμετέχουν χώρες μέλη, περιφέρειες, αλλά και το ευρωπαϊκό επίπεδο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο μηχανισμός αυτός βέβαια πρέπει να υιοθετηθεί από όλε τις χώρες μέλη για να είναι και αποτελεσματικός. Δηλαδή θα ισχύει η νομοθεσία και οι ρυθμίσεις της μιας χώρας και στην άλλη χώρα όσο κρατάει η διεκπαιρέωση του έργου. Πρώτα απ' όλα θέλω να υπογραμμίσω όμως ότι ο μηχανισμός αυτός είναι προαιρετικός σε θελοντική βάση. Έτσι καθισχάζονται κάποιες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί όσον αφορά την αναλλαγικότητα και την, επικουρικότητα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται λοιπόν για προαιρετική εφαρμογή. Τώρα από πλευρά των χωρών μελών έχουν ε, διάφορες δυνατότητες οι χώρες μέλη για να συμμετέχουν. Πρώτα απ' όλα προτείνει τον μηχανισμό προαιρετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως είπαμε. Άπαξ και μία χώρα. Συγγνώμη, λέει ο Επιτροπός. Η πρόταση έχει ως εξής. Ας σκεφτούμε τις χώρες Μπενελούξ που έχουν διασυνοριακές περιοχές και θέλουν να διεκπερώσουν ένα έργο πιο εύκολα εφόσον ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις σε όλες τις χώρες. Αν δεν υπάρχει ήδη ένας τέτοιος μηχανισμός, τότε πρέπει, αναγκάζεται δηλαδή η χώρα, κάθε χώρα μέλος, να επιλέξει αυτόν τον ευρωπαϊκό διασυνορικό μηχανισμό. Αλλά τότε πώς πρόκειται για προαιρετική λύση, θα μου πείτε. Και πού πάει η επικουρικότητα. Γι' αυτό όμως υπάρχουν τα άρθρα 1 και 4 που λένε ότι η χώρα μέλος μπορεί να διαλέξει είτε έναν τέτοιο μηχανισμό, είτε έναν μηχανισμό που ήδη υπάρχει, είτε να αποφασίσει για έναν νέο μηχανισμό, καινούριο. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή. Ούτε είναι υποχρεωτικό άπαξ και έχει αποφασίσει μια φορά να ακολουθήσει τον Ευρωπαϊκό Διασυνορικό Μηχανισμό ότι θα το κάνει πάντα. Είναι για ένα συγκεκριμένο έργο. Πρέπει σε θελοντική βάση, όπως είπαμε, να αποφασίζουν οι χώρες και οι περιφέρειες και όχι να γίνει υποχρεωτικός. Βέβαια, πρέπει όλες οι χώρες να διαθέτουν ένα διασυνοριακό σημείο συντονισμού που να συντονίζει τα πράγματα. Και αυτός ο διασυνοριακός ε, κόμβος, αυτό το διασυνοριακό σημείο συντονισμού να υπάρχει σε κάθε χώρα. Δηλαδή θα υπάρχει στο Λουξεμβούργο, αλλά θα συντονίζεται και με το αντίστοιχο σημείο διασυνοριακού συντονισμού στην γείτονα χώρα. Και καθήκον τους είναι να δούνε σε τι βαθμό ταιριάζει η κάθε λύση. Υπάρχει βέβαια και η εδαφική συνεργασία. Εδώ μπορεί να είναι αλακάρτη λύση, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε χώρας και της κάθε περιφέρειας. Η μία χώρα υιοθετεί τις ρυθμίσεις της γείτονος χώρας, σε θελοντική βάση. Άρα σεβόμαστε την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Για το θέμα του πόσο είναι υποχρεωτικός ή όχι, ε, είπαμε, είναι θελοντικός και στη θεωρία αλλά και στην πράξη γιατί εξηγήσαμε ότι έχει κάθε φορά τη δυνατότητα κάθε χώρα να επιλέξει κάποια άλλη λύση. Υπάρχουν τα άρθρα 10, 12 και 16 που μιλούν για μια χρονική διάρκεια τριών με έξι μηνών. Σίγουρα χρειάζονται νομικές προδιαγραφές για να αποφεύγονται όλα τα εμπόδια και ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις της μιας χώρας στην γείτονα χώρα. Έχει λοιπόν ένα χρονικό διάστημα στη διάθεσή της η κάθε χώρα, αλλά κάποια στιγμή βέβαια θα πρέπει να καταλήξει και να αποφασίζει αν θα δεχτεί αυτή τη ρύθμιση ή όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συμπεριλάβει υποδομές και έργα τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν, ακόμα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτήν τη ρύθμιση, σε αυτό το μηχανισμό. Έχουμε υποδομές από τη μία και υπηρεσίες οικονομικού ενδιαφέροντος από την άλλη. Αυτό είναι ο ορισμός. Πρέπει βέβαια να δοκιμαστεί πρώτα ο μηχανισμός για να δούμε κατά πόσο στην πράξη όντως αποτελεί μια λύση ή όχι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής ευθύς εξ αρχής. Ελπίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια ισορροπημένη ρύθμιση. Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση διασυνοριακών προβλημάτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και γι' αυτό φτιάξαμε το Ίντερεκ, γι' αυτό έχουμε φτιάξει και τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας και τώρα έχουμε και αυτόν τον μηχανισμό. Πρέπει να είναι αποτελεσματικό ο μηχανισμό. Όποιο και, αν είναι ο μηχανισμός που επιλέγουν οι χώρες, έτσι ώστε να μπορούν οι παραμεθόριες περιοχές να χαίρουν ευημερίε, να συνεργάζονται και να έχουν οικονομική ανάπτυξη. Είχα πει ότι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια ακρόαση. 10 με 1,5. Υπάρχει, οργανώθηκε αυτή η ακρόαση και εννοείται ότι είσαστε όλοι προσκεκλημένοι και κυρίως βέβαια οι σκιώδεις εισηγητές. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές, μέλη Επιτροπής ε, Ρέγγι και να σας ενημερώσω ότι ο εισηγητής από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή είναι εδώ και είναι έτοιμος να μας παρουσιάσει την γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ. Επομένως, να ξεκινήσουμε με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Ε, κύριε Τσέλερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ και τον συνάδελφο Φαν Μίλτεμπουργκ, τον εισηγητή μας ε, για μια πολύ περιεκτική δουλειά που έχει ήδη κάνει οι διαστημικές περιφέρειε των 40% τη ε, ε, επικράτησης ένωσης, το 1 τρίτο των πολιτών, οι διάφορε υποδομέ. ε, Πολλές φορές όμως υπολείπονται σε αυτές τις παραμεθόρες περιοχές και υπάρχουν δυσκολίες ε, για διασυνοριακές συνδέσεις. Ε, παραδειγματικά το, το παρελθόν ε, πολλές φορές ήταν και πρόσφορο έδαφος περιοχές αυτές για διαφόρους πολέμους κτλ. Τώρα το θέμα είναι ότι η συνεργασία είναι το ζητούμενο για την κοινωνική και οικονομική συνοχή, αλλά υπάρχει και εδαφική συνοχή και κυρίως πρέπει να προσέξουμε εδώ τις διασυνοριακές ε, περιφέρειες. Έχουμε ήδη τη δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg και στην προηγούμενη περίοδο, στην προηγούμενη θητεία, ε, είχαμε ε, ακόμη περισσότερη πρόοδο στον τομέα της συνεργασίας, όμως στην πράξη βλέπουμε ότι στις διασυνοριακές αυτές περιφέρειες εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια και υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών που δεν συνεργάζονται επαρκώς. Επομένως δημιουργούνται προβλήματα αντί να δημιουργούνται να έχουμε βελτιώσεις. Ε, το 2014 ε, η Προεδρία του Συμβουλίου ανέπτυξε την πρωτοβουλία ε, της δημιουργίας ενός μηχανισμού όπως τον λέμε τώρα ε, να συμπληρωθεί η όλη δηλαδή ε, διασυνορική συνεργασία με αυτό τον Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Μηχανισμό. Έχουμε λοιπόν τώρα αυτή την πρόταση και θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπήκε σε αυτή την προσπάθεια να ε, δρομολογήσει αυτό τον μηχανισμό, τον Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Μηχανισμό. Ε, υπάρχουν ε, αντιδράσεις ε, βέβαια και σε σχέση με τα κράτη-μέλη και κάποια ομοσπονδιακά κρατήδια της Γερμανίας επίσης διαμαρτύρονται ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας της επικουρικότητας, ότι μπορούν να χάσουν κάποιες αρμοδιότητες. Πάντως, σε ό,τι αφορά την ε, παραμεθόρια συνεργασία, νομίζω ότι ε, οι σημερινοί μηχανισμοί δεν την εγγυώνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, άρα υπάρχουν ανάγκες και γι' αυτό χαιρετίζω την πρόταση όπως έχει κατατεθεί και πιστεύω ότι και με την ε, συζήτηση που θα ακολουθήσει θα βελτιωθεί αυτή η πρόταση έχει διατυπώσει συγκεκριμένε άλλωστε προτάσει και ο εισηγητή Φαν Μίλτεμπουργκ σε ό,τι αφορά παραδείγματο χάρη ε, το προαιρετικό, τον εθελοντικό χαρακτήρα. Θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν κάποια ελευθερία στα στις περιφέρειες ή στα ε, ομοσπονδιακά κρατήδια ενίοτε, αλλά πρέπει να υπάρχει και κάποιος έλεγχος όταν χρειάζεται. Να, υπάρχουν και κάποια, να υπάρχει και ένας υποχρεωτικός χαρακτήρας δηλαδή εκεί που χρειάζεται για να μπορέσει να λειτουργήσει καλά η συνεργασία που έχει άμεση σύνδεση και με την ε, συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν προτάσεις Αν δούμε τον μέχρι τώρα εφιστάμενο μηχανισμό, ε, το Ιντερεκ, τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Αδαφικής Συνεργασίας, υπάρχουν ε, ε, ανάγκες να υπάρχει συμπληρωματικότητα και όχι το ένα ε, μηχανισμός να είναι αντίθετος στον άλλον, με τον άλλον και να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Φαντάζομαι ότι μπορούμε σε κάποια σημεία να διατυπώσουμε με πιο ακριβή τρόπο, με βελτιωμένο τρόπο την νομοδότηση. Παραδείγματο χάρη δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια, τα σύνορα μην είναι εμπόδιο, ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τις ε, διασυνοριακές περιφέρειες ε, που ε, προσπαθούν να προωθήσουν κοινά σχέδια. Το ίδιο ισχύει και για τις υπερπόντιες χώρες και εδάφια, αν θέλουν και αυτές να συμμετέχουν. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε με κάποιες τροπολογίες το οποίο και θα κάνουμε. Ελπίζω πάντως ο νέος αυτός μηχανισμός να εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία. Ε, πρέπει να σκεφτούμε τις ανάγκες αυτών των διασυνοριακών περιφερειών. Δεν είναι ακριβώς ε, το ίδιο. Ε, πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Ε, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ότι στην υπηρετική Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά θα πρέπει να τα προωθήσουμε. Ευχαριστώ. Πρώτα, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τσέλερ. Θα δώσω... Και τώρα το λόγο κύριος Χάουρτ. Σκιώδης, ηγητής, παρακαλώ. Όντως, Πρόεδρε, σκιώδης είμαι και ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να εκπροσωπήσω την κυρία Σμόλκοβα. Ξεκινώ λοιπόν ευχαριστώντας τον εισηγητή, κύριο Φανούντελμπεργκ, για το είναι πολύ καλά στοιχειοθετημένη έκθεση, το σχέδιο εκθέσεως είναι ευπρόσδεκτος ο μηχανισμό όπω έχω ήδη δηλώσει, και θα ήθελα να τεθεί σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατό. Θετικό λοιπόν κρίνω το ότι μπορούμε να οργανώσουμε την ακρόαση του συναδέλφου ε, την κατάλληλη στιγμή. Θα ήταν χρήσιμο πιστεύω να διευρυνθεί το πεδίο της έκθεσης σε διάφορα σημεία και πτυχές ο ρόλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραδείγματι, περισσότερε προσπάθειε πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία και τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ, οι οποίε θα πρέπει και περισσότερε πληροφορίε να λαμβάνουν μέσω ειδική ε, στρατηγική επικοινωνία, παραδείγματι, για να αντιλαμβάνονται καλύτερα τα πλεονεκτήματα ενό τέτοιου μηχανισμού και να ικανοποιούν τους στόχους του. Επιπλέον, στην υλοποίηση του μηχανισμού, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να ε, προσφέρουν τη γνώμη τους, να γίνεται διαβούλευση δηλαδή, μαζί τους, τακτικά. Μια μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση στη διαδικασία της ε, εφαρμογής έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μια πενταετής περίοδος αξιολόγησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μου φαίνεται ικανοποιητική. Ο ορισμός των έργων και το πεδίο του μηχανισμού θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε στην πρόταση με έργα υποδομής και υπηρεσίες γενικής, γενικού συμφέροντος. Ωστόσο, ε, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στις διατάσεις μας, συνεργασία για τις υπηρεσίες τη ανάγκη, σε παραδείγματι, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, ε, μεγάλων ατυχημάτων κτλ. Αντιλαμβάνομαι ότι ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να έχει πολλές δυσκολίες σε διοικητικό επίπεδο, αλλά θεωρώ πως ε, και η επικοινωνία με τους φορείς ε, εξ αρχής θα μπορούσε να περιορίσει τις οποίες δυσκολίες. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε και να περιορίσουμε τις ε, συνέπειες ε, και τις δυσκολίες προς όφελος όλων των πλευρών. Προσβλέπω στην περαιτέρω συζήτηση και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όζοκ. Αν προσφέρω καλά το όνομά σας, με συγχωρείτε λέει η Πρόεδρος. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώ εδώ τον συνάδελφο κύριο Πιοτρόφσκι και θα περιοριστώ στην ανάγνωση της δικής του τοποθέτησης. Ως και ηγητής υποστηρίζω την ιδέα για την κατάργηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα του μηχανισμού όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο έκθεσης του συναδέλφου ε, οδηγεί προς την κατεύθυνση αυτή που είναι και σωστή πιστεύω, ωστόσο με μία επιφύλαξη σχετική με την ε, τροπολογία υπαριθμών 10 καθώς φρονώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ε, διακριτικό περιθώριο για, τον, για, την κατάρ, για τη σύσταση των εθνικών συντονιστικών τους αρχών. Διαφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής για μια τόσο χρονοβόρα διαδικασία προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός δεν θα είναι χρήσιμη για εκείνους που αναπτύσσουν διασυνοριακά έργα και η εφαρμογή νομοθεσίας του ενός κράτους μέλους στην επικράτεια ενός άλλου ε, μας γεννά πολύ σοβαρές ανησυχίες και αμφιβολίες προς τα νομικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του κυρίου Παπαδημούλη παρακαλώ. Όχι, εκ μέρους του κ. Ροπέ. Κύριε Ντεμάτο παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ πάνω απ πρώτα απ' όλα τον συνάδελφο για το, η του σχεδίου πρότασης ε, εκθέσεως. Ε, συζητούμε πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια τους μηχανισμούς που χρειάζονται για να γίνει πιο απτή ε, για τον πολίτη, να έρθει πιο κοντά στις ανάγκες του και να γίνει και πιο ελαφριά σε όρους διοικητικού άχθους η διαδικασία για τις περιφέρειες. Οι προτάσεις ακολουθούν το σωστό δρόμο, παρότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που δεν είναι ακόμη σαφή και που βλέπω ότι και ο ίδιος ο συνάδελφος επισημαίνει με κάποιες τροπολογίες του. Έχουμε μια διαδικασία λοιπόν που έχει κρατήσει δύο χρόνια και με στοιχεία που έχει συλλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί δύο χρόνια αρκετά ανησυχητικά. Οι παραμεθόριες περιοχές εν γέννη δηλαδή φαίνεται να έχουν κατώτερα οικονομικά αποτελέσματα και επιδόσεις σε σχέση με τις περιοχές που βρίσκονται στην ενδοχώρα των κρατών μελών. Είτε πρόκειται για νοσοκομεία, πανεπιστήμια ή άλλες υπηρεσίες. Βλέπουμε ότι είναι λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες στα παραμεθόριες περιοχές και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το κέντρο δυνατό και με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό και το πλαίσιο μέσα στο οποίο συζητούμε σημαίνει μέτρα τα οποία θα ξεπερούν την απλή οικονομική ενίσχυση από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα την ε, καθιστά πολύ πιο απτή για τις παραμεθόριες περιοχές, γιατί εκεί τα προβλήματα δεν μπορούν να επιληθούν μόνο με το Interreg, δηλαδή με τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης. Έχουμε να κάνουμε επίσης με, μια, με την ανάγκη να συμπληρωθεί όχι μόνο η οικονομική ενίσχυση του πλαισίου του Interreg, αλλά ταυτόχρονα και να προσφερθεί πολιτική υποστήριξη, όπως σε παραδείγματι με, τις ευρωπαϊκές, με τους ευρωπαϊκούς φορείς διασυνοριακής ε, που όμως δεν έχουν νομικά τη δυνατότητα να ε, εισαγάγουν νομοθεσία. Άρα πρέπει να, ξεπερα... να υπερβληθούν οι νομικοί περιορισμοί. Ο μηχανισμός ε, που προβλέπεται είναι ε, προαιρετικό. Ε, εδώ βλέπουμε μια τροπολογία του εισηγητή όπου η διατύπω, που επισημαίνεται ότι η διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γεννά αρκετές ανησυχίες. Δηλαδή ένα κράτος μέλος φαίνεται θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ένα μηχανισμό για οποιοδήποτε διμερές ή πολυμερές σχέδιο ή θα μπορούσε να ε, επιλέξει διαφορετικούς δρόμους για τα έργα σε παραμεθορίες περιοχές. Ε, τα κράτη-μέλη που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τους κατάλληλους μηχανισμούς όμως φαίνεται να μην έχουν επιλογή παρά μόνο της καταφυγής στον διασυνοριακό ευρωπαϊκό μηχανισμό. Άρα θα πρέπει, επαναλαμβάνω, η συνεργασία να γίνεται σε, σε, με όρους προαιρετικούς και κατά περίπτωση ένα κράτος μέλος με βάση ε, διατυπώσεις μεταβλητή γεωμετρία και έτσι τα κράτη-μέλη τα οποία εντοπίζουν ένα νομικό εμπόδιο σε διασυνοριακό επίπεδο θα μπορούν να επιλέξουν αν θα χρησιμοποιήσουν έναν εφιστάμενο μηχανισμό ή αν θα εισαγάγουν έναν νέο μηχανισμό ή αν θα επιλέγουν τον διευρωπαϊκό μηχανισμό. Και έτσι για λόγους ε, βέβαια που θα εξηγούνται ε, με την κατάλληλη αιτιολογία θα μπορούν να ε, αποδιαρθρώνουν εμπόδια διοικητικά ή νομικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπρέσσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους για τη φωνή μου. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο. Με μεγάλη προσοχή άκουσα την ε, τεκμήριωσή του. Οφείλω όμω να πω πω ε, βρίσκομαι σε αμηχανία, γιατί μιλούμε για πρόταση κανονισμού και όχι οδηγία. Το πλεονέκτημα που προσφέρει ένα κανονισμό σε μια τέτοια περίπτωση, ένα τέτοιο υλικό, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το έχουμε παληθεύσει με το JECT, το, την Ευρωπαϊκή Ομάδα δηλαδή Δαφικής Συνεργασίας ε, και γι' αυτό έχει επιλεγεί η μορφή του κανονισμού και δίνει βέβαια κάποια περιθώρια ελευθερίας κινήσεων, αλλά διαπιστώνεται ότι αυτά τα περιθώρια σε πολλές περιπτώσεις δεν τα έχουν εφαρμόσει τα κράτη-μέλη, με αποτέλεσμα πολλές δυσκολίες για τις παραμεθόριες ε, περιοχές. Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι δεν μιλούμε για μικρά κράτη μόνο, μιλούμε και για μεγάλα κράτη, των οποίων οι... Ε, πρωτεύουσε μπορεί να βρίσκονται στο κέντρο τη ενδοχώρα και να μην έχουν κανένα πρόβλημα διασυνοριακή συνεργασία και εκ τούτου να μην ενδιαφέρονται καθόλου ή να παραγνωρίζουν τι δυσκολίε ω προ την συνεργασία σε διασυνοριακό επίπεδο. Και γι' αυτό και η συνάδελφο νωρίτερα, κυρία Νταμάτο, μίλησε για τι δυσκολίε ιδιαίτερα των παραμεθωρίων περιοχών που έχουν χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξη και λόγω τη αδυναμία συνεργασία μεταξύ του. Ε, παρακαλώ λοιπόν τον συνάδελφο εισηγητή να παρακολουθήσει με προσοχή και να κοιτάξει την προσαρμογή και των τροπολογιών και προτάσεών του, γιατί πρέπει νομίζω να επαγρυπνούμε ώστε να μην ε, καταστεί απολύτω περιπτωσιολογική αυτή η λύση του κανονισμού. Δεν μπορεί να είναι περιπτωσιολογικό εδώ τα κράτη-μέλη σε όρου προαιρετικού και προφανώ κατόπιν αιτήματο τη σχετική της ε, περιφέρειας της παραμεθόριας δίνανται ακόμα και να αποφασίσουν με ποια μέσα θα διευκολύνουν τη συνεργασία. Εάν αυτό γίνει περιπτωσιολογικά, κατά περίπτωση. Νομίζω ότι ο καθένας που έχει ασχοληθεί με τα περιφερειακά θέματα ε, ή την τοπική συνεργασία δεν θα ξέρει ότι αυτό θα κρατάει μήνες αν όχι χρόνια γιατί κάθε φορά θα πρέπει να κρίνονται οι διάφορες συνθήκες κατά περίπτωση. Θα επιδεινώνεται λοιπόν το περίπλοκο της, ε, του εγχειρήματο και δεν θα διευκολύνεται. Άρα θα καταστεί ανέφικτο όλο αυτό το εγχείρημα και παρακαλώ τον συντάκτη, τον ε, εισηγητή αλλά και τους συναδέλφους και οδησηγητές ε, να μην λησμονούμε ότι πρόκειται για έναν κανονισμό, ένα νομοθέτημα ασφαλές και άμεσης εφαρμογής το οποίο εξασφαλίζει για τον Ευρωπαίο πολίτη και άρα και τις περιφέρειες ε, την ασφάλεια της άμεσης εφαρμογής και άρα διευκολύνει έτσι τη διασυνοριακή συνεργασία. Οι περιφέρειες, οι τοπικές αρχές δεν βλέπουν να αναγνωρίζεται ο ρόλος τους και πάνω απ' όλα να διευκολύνεται η ταχεία εφαρμογή αυτών των δυνατοτήτων συνεργασίας από πλευρά των κρατών. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ποιος άλλος? Ο κύριος Φανής Λερόι. Ναι, σύντομα. Και στα... στα Ολλανδικά. Την προηγούμενη φορά επίσης είχαμε συζητήσει μεταξύ μας για τον μηχανισμό τον προηγούμενο, του ευρωπαϊκού Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας και τώρα λέγαμε ότι θα μπορούσαν έτσι να μεταφέρουν μέρος των αρμοδιοτήτων του σε αυτόν τον μηχανισμό. Αρκεί να το αναγνωρίσουν βέβαια οι χώρες μέλη, οι εκπρόσωποι των αρχών. Και να μην γίνεται αυτό κατά περίπτωση, αλλά είναι κάτι μόνιμο. Από την άλλη μεριά βρίσκω πάρα πολύ καλό που η εισηγητής λέει ότι παραμένει σε προαιρετική βάση. Και μπορεί να αλλάζει το πράγμα από χώρα σε χώρα. Άλλος να τον χρησιμοποιεί πιο πολύ, άλλος πιο λίγο. Μίλησε à la Να προχωρήσει αυτός ο μηχανισμός. Ωραία. Προσοχή όμως. Τι είναι τελικά αυτό που προσθέτει αυτός ο μηχανισμός. Ο προηγούμενος τι ήταν πολύ δύσκολος. Γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη λύση. Αυτά. Πρόεδρο. Σε ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπάρατ, ο οποίος ε, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής. Κύριε Μπάρατ, έχετε εσείς το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μπορώ να μιλήσω ουγγρικά. Μπορώ μάλιστα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους της Οπλής Κοινωνικής Επιτροπής για την πρόσκληση Μπορεί να μην φαίνεται εκ πρώτη όψεω τόσο σημαντικό αυτό ε, ο κανονισμό, όμω ε, όπω είπαν και ε, βουλευτέ, θα λύσει πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Και οι λύσει αυτέ θα μα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο κοινό μέλλον. Επομένω, είναι σημαντικό αυτό ο μηχανισμό. Από ιστορική πλευρά, τα σύνορα, οι μεθορικές περιοχές ε, έπαιζαν πάντοτε ένα σημαντικό ρόλο. Ε, δεν είναι ίδια η κατάσταση ε, όπως παλαιότερα, αλλά σίγουρα τα σύνορα υπάρχουν και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Υπάρχει και μία μελέτη που λέει ότι αν δεν υπήρχαν σύνορα θα αυξανόταν το έπτον των περιοχών των παραμεθόριων και κατά 8%. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι ε, στην ε, άρση των συνόρων, ε, με την αρσοστό θα αποδεσμευθεί ένα τεράστιο αναπτυξιακό δυναμικό. Και βέβαια θα προωθηθούν και θα ωφεληθούν τομεί όπω η παιδεία, η υγεία κτλ. Πάρα πολλέ ακροάσει έχουν οργανωθεί. Θα ήθελα να σας μιλήσω για δύο συγκεκριμένα περιπτώσεις ε, σε μια μικρή πόλη στην Ολλανδία ξέσπασε μια μεγάλη πυρκαγιά και δεν μπορούσαν να πάνε Γερμανοί πυροσβέστες γιατί αυτό ήταν απαγορευμένο. Χρειαζόντουσαν άδειε, εγκρίσει κτλ. Ή στο Στρασβούργο, για παράδειγμα, υπάρχει ένα σχολείο ε, που δεν έχει πισίνα. Ο δάσκαλος με τα παιδιά από τη Γαλλία πηγαίνει στη Γερμανία ε, μπορεί να, να πάει ε, στην ε, πισίνα, αλλά πρέπει να πάρει κάποια συγκρίση από την Γερμανία κτλ. Ε, όπως, όπως αυτά καταλαβαίνετε ότι περιπλέκουν την κατάσταση αχρίαστα. Στον κανονισμό λοιπόν αυτό γίνεται λόγος και για την αρχή της επικουρικότητας. Είναι σημαντικό να υπάρχει επικουρικότητα και Σίγουρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, ε, τον προαιρετικό χαρακτήρα. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να είναι προαιρετικός. Θα μπορούν οι τοπικές αρχές να αποφασίσουν κατά πόσο να επιθυμούν να συμμετέχουν ή όχι. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί. Και αυτό το οποίο προτείνουμε επίσης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει την παρακολούθηση, τον έλεγχο να αναλύει δηλαδή τις διαδικασίες, ε, να κάνει κάποια έρευνα και έπειτα να προωθεί ε, τις, κοινέ, τις ε, καλές πρακτικές. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι πολύπλοκη εφαρμογή, ενδεχομένως να είναι, πάντως πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώ δεν υπάρχει κάποια αναπτυξιακή στρατηγική ακόμη για το πώ θα μπορούσαν να ενταχθούν αυτοί οι μηχανισμοί σε μια στρατηγική. Έχουμε τη στρατηγική ε, αναπτυξιακή που δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως. Γίνεται λόγος για τις μακροπεριφέρειες, τη μακροπεριφερειακή συνεργασία, αλλά δεν γίνεται λόγος για το μέλλον ε, των ε, της παραμεθοριακής, της δεσυνοριακής συνεργασίας. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα ε, που δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί από μια τέτοια συνεργασία. Επίση, πολύ σημαντικό είναι ο συντονισμό. Ε, θα πρέπει επίση ε, χρηματοδότηση να εξασφαλίσει και θα πρέπει να υπάρχει και επικοινωνία, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλε αυτέ οι προτάσει, αυτέ οι λύσει. πρέπει να ωφελήσουν τους πολίτες, πρέπει να ωφελήσουν τις περιφέρειες. Αυτό θα συμβεί μόνο αν υπάρχει σωστή επικοινωνία και δημοσιοποίηση αυτών των πρωτοβουλίων. Πολλέ φορέ ε, αποτυγχάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες επειδή δεν υπάρχει επαρκή ε, προβολή τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την πρόσκληση. Και ελπίζω να ε, προχωρήσει πολύ καλά η διαδικασία αυτή. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχετε κύριε Φαμπρέσκα πολυπληθή ομάδα εδώ βλέπω, άρα μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Όντως. Τέσσερις παρατηρήσεις καταρχήν. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα πολύ τον εισηγητή για την θετική του αντιμετώπιση και την οικοδομητική του έκθεση. Για κάποια ζητήματα όμως έχουμε κάποιες ανησυχίες. Τρία-τέσσερα. Λοιπόν, το πρώτο και τέθηκε εδώ στη συζήτηση είναι ότι μας απασχολεί το ότι υπογραμμίζεται τόσο πολύ ο προαιρετικός χαρακτήρας. Και μάλιστα υπογραμμίζεται ξανά και ξανά στις τροπολογίες. Εμείς φοβούμεθα ότι θα είναι τόσο προαιρετικός τελικό μηχανισμός αυτός που δεν θα χρησιμοποιείται καθόλου. Και δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει, δεν είναι προς το συμφέρον μας. Δεύτερον, έχουμε κάποιες δυσκολίες να κατανοήσουμε πώς ακριβώς ένας τέτοιος μηχανισμός θα δημιουργείται για μεμονωμένα έργα και θα διαλύεται αμέσως μετά και μετά από λίγα χρόνια ίσως ξαναδημιουργείται. Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι. Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι ένας μηχανισμός ε, με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται τα νομικά ζητήματα, τα διασυνοριακά, και όχι ένα εργαλείο το οποίο θα ενεργοποιείται όσο υπάρχει ένα έργο και θα πανεργοποιείται αμέσως μετά. Το θέμα τώρα που τέθηκε το κατά πόσο είναι μια νέα μορφή ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας δεν θελήσαμε να δημιουργήσουμε εδώ ένα νέο νομικό πρόσωπο. Δεύτερη ανησυχία. Βεβαίως και σημειώνουμε ότι θα μπορούσε κανείς να αναπτύξει και άλλους αποτελεσματικούς μηχανισμούς ή εργαλεία. Όμως, στη δικιά μας τη σύσταση, η ιδέα είναι ότι εφόσον υπάρχει διαθέσιμος ένας ευρωπαϊκός διασυνοριακός μηχανισμός, γιατί να σπαταλήσει μια χώρα, μια περιφέρεια, θέα ουσία, δυνάμεις, ε, χρήματα κτλ. για να δημιουργήσει κάποιον άλλον μηχανισμό. Επίσης θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι φυσικά και θέλουμε να ελέγξουμε κατά πόσο μια τέτοια αναλλακτική λύση, ένα τέτοιο μηχανισμός επιτυχάνει τους ίδιους στόχου, δηλαδή να ξεπεραστούν τα νομικά εμπόδια ή όχι όντως πρέπει να υπάρχουν ε, κριτήρια όσον αφορά τις προθεσμίες, το συντονισμό κτλ. που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε αν είναι μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση αυτός ο μηχανισμός. Και τέλος, ε, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ασυνέπειες εδώ. Γιατί διαβάζοντας την έκθεσή σας, αν καταλαβαίνουμε καλά, λέει ότι όλες οι χώρες μέλη πρέπει να διαθέτουν ένα διασυνοριακό σημείο συντονισμού. Αλλά τότε γιατί να έχει εναλλακτικού μηχανισμούς. Δηλαδή, αν βάσει της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας, βάσει αυτού του κανονισμού είναι υποχρεωμένες όλες οι χώρες να έχουν ένα διασυνοριακό σημείο συντονισμού, γιατί συγχρόνω να μπορεί να ακολουθήσει άλλε εναλλακτικέ λύσεις και μηχανισμούς. Δηλαδή, μα φαίνεται ότι υπάρχει κάποια συνέπεια εδώ μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Άλλο θέμα, διευκρινιστικά. Στην έκθεση αναφέρονται συχνά κοινά προγράμματα, ενώ το άρθρο 2 του σχεδίου κανονισμού που αναφέρεται στον ορισμό των κοινών έργων δεν τροποποιείται. Οπότε η ερώτησή μας είναι, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλάμε για έργα που είναι υποδομής διασυνοριακά, αλλά και υπηρεσιών κοινοφελού ενδιαφέροντο διασυνοριακά. Οπότε η ερώτησή μας είναι οι τροποποίησεις που προτείνονται έχουν να κάνουν μόνο με συγκεκριμένα κοινά έργα ή καλύπτουν και τις δύο πτυχές. Εμείς δεν βλέπουμε στην πράξη πώς μπορούν να γίνουν αυτές οι τροποποίησεις. Και τέλος για τις προθεσμίες. Σημειώνουμε ότι κάθε προθεσμία για τις χώρες μέλη και ισχύει και στο Συμβούλιο το ίδιο, φαίνεται να παρατείνεται. Ενώ οι προθεσμίες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επιβραδύνονται. Δηλαδή πρέπει να αντιδράει πιο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ οι χώρες μέλη έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους. Και η είπε ότι τόσο μικρές προθεσμίες για τις διαδικασίες έχουν σαν στόχο να προστατεύσουν τους τοπικούς φορείς. Οι τοπικοί φορείς πιστεύουμε και εμείς ότι πρέπει να αποφελούνται από σύντομες προθεσμίες ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι οι επαφές τους με τις εθνικές αρχές πρέπει να γίνονται μέσα σε πιο περιορισμένα πλαίσια. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ ευχαριστούμε. Κύριε Βαν Μίλτεμπερ, για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στους συναδέρφους. Πρώτα απ' όλα, στον κύριο Τσέλερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε τι γίνεται με τις τρίτες χώρες. Ε, σωστά. Νομικά είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός. Έτσι. Οπότε δεν μπορεί να δεσμεύσει κανέναν εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε και το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Brexit. Κύριε Μπρέσο, είπατε ότι πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, ώστε να μην είμαστε υπερβολικά απαιτητικοί. Και αυτό λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ όμως σκέφτομαι ότι έτσι κι αλλιώς πρέπει και βάσει της πρότασης της Επιτροπής κάθε φορά πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο οι κανόνες τηρούνται όπως πρέπει και στη χώρα Α και στη χώρα Β και να δούμε κατά πόσο προκύπτουν ή δεν προκύπτουν νομικά ζητήματα και πώς αυτά επιλύονται. Οπότε κάθε φορά θα πρέπει να δούμε πολύ καλά ποιες είναι οι λύσεις που προσφέρονται στα νομικά εμπόδια και στις νομικές δυσκολίες. Πρόκειται μια, για μια ολόκληρη διαδικασία βέβαια που περιλαμβάνει ο μηχανισμός. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά βέβαια αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που λέει ότι είναι καλύτερα μια φορά να καθεδρύεται αυτός ο μηχανισμός, μα έτσι κι αλλιώς οι ε, αποφάσεις και οι αξιολογήσεις θα γίνονται κατά περίπτωση, για κάθε έργο. Ο άλλος προβληματισμός είναι το προαιρετικό. Μα έχουν τεθεί ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επικορικότητα και την αναλογικότητα και από το Cambridge University. Πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά τι απάντηση θα δίνουμε και πιστεύουμε ότι με τον προερωτικό χαρακτήρα μπορούμε να καθισκάσουμε τις ανησυχίες των χωρών μελών. Καλύτερα να ξεκινήσουμε με ένα τέτοιο κανονισμό που προτείνουμε στις χώρες σε θελοντική βάση είναι ένα καλό βήμα προς τη σωτή κατεύθυνση και μετά θα δούμε, όπως λέω και εγώ μετά από τρία χρόνια θα αξιολογήσουμε την κατάσταση, θα δούμε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και ανάλογα θα προσαρμόσουμε τη ρύθμιση αυτή. Ίσως γίνει περισσότερο υποχρεωτικός αυτός ο μηχανισμός, δεν ξέρω. Αν δούμε ότι πολλές χώρες το θέλουν, ναι. Τώρα για αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα συγκεκριμένα έργα, το σημείο 2 που αναφέρεται στους ορισμούς, λέει ότι κάθε φορά που υπάρχει ένα κοινό έργο Αυτό ισχύει. Και τέλος, η προθεσμία. Τρεις μήνες φαίνεται καλό, αλλά νομίζω ότι για ορισμένες περιπτώσεις και για ορισμένες χώρες, αν τον Ιούνιο, αν τον Ιούνιο για παράδειγμα, τεθεί ένα νομικό ζήτημα και έχουμε μετά το καλοκαίρι τις διακοπές και πούμε τρεις μήνες, δύσκολα θα πάρει κανείς σοβαρή απάντηση. όταν πρόκειται για περίοδο διακοπών, θα έπρεπε τρει μήνε να γίνονται έξι. Ξέρω πολύ καλά τα νομικά ζητήματα, πόσο δύσκολα λύνονται σε επίπεδο Υπουργείων. Τρει μήνε στη χώρα μου μου φαίνεται ότι δεν φτάνει. Γιατί πολλά ζητήματα πρέπει να περάσουν από πολλά Υπουργεία και ακόμα και μέσα σε ένα Υπουργείο από πολλές υπηρεσίες. Οπότε οι τρεις μήνες δεν θα φτάνουν. Εγώ προτιμάω να είμαστε ρεαλιστές και να κρατήσουμε τους έξι μήνες. Καλύτερα να βρούμε μια καλή λύση και ας κρατά έξι μήνες. Αυτά. Κατά τα άλλα προσβλέπω σε καλή συνεργασία με τους σκιώδεις συζητητές και θέλω να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για την στήριξή της και γενικότερα τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη νομική υπηρεσία που με βοήθησαν πολύ για κάτι που φαίνεται μια εύκολη πρόταση έτσι από πρώτο χέρι, αλλά επειδή πρόκειται για νομικά ζητήματα είναι πολύ πιο περίπλοκη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φαν Μίλτεμπουργκ. Προθέσουμε κατάθεση τροπολογιών. Προτείνω να είναι 22 Οκτωβρίου 6 ώρα το απόγευμα. 22 Οκτωβρίου 6 ώρα το απόγευμα. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο της μερσιάς διάταξης τώρα. Εξέταση σχεδίου έκθεσης σε ό,τι αφορά την νομοθετική πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής. Η συγητής μας είναι ο κύριος Κοτσολίνο και είναι έτοιμος να μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του. Θέλω απλά να σας πενθυμίσω πως πρόκειται για ένα από τα νομοθετικά ζητήματα που άπτονται και του σε σε πλαισίου έχουν μεγάλη σημασία για εμάς, τα θέματα αυτού του φακέλου. Είχαμε συζήτηση, είχαμε ανταλλαγή απόψεων στις 3 Σεπτεμβρίου εδώ στην Επιτροπή μας. Σήμερα θα ακούσουμε τον κύριο Κοτσολίνο να μας παρουσιάσει την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεσή του. Ήδη ε, περιλαμβάνει 72 τροπολογίες στην πρόταση της Κομισιόν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Κοτσολίνο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Αναφέρθηκε και νωρίτερα ότι έχουμε να κάνουμε 72 τροπολογίες, 44 αφορούν το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, είμαστε όμως μόλις στην αρχή της πρότασης και διατεθειμένοι φυσικά να ε, συλλέξουμε τις προτάσεις των συναδέλφων σκιωδών συγητών. Μια δουλειά που τους άλλους μαζί θα κάνουμε από κοινού στην Επιτροπή μας. Ξεκινώ με τις εξής ε, δύο προκαταρκτικές τοποθετήσεις ότι η συνείδηση πως ε, έχουμε να κάνουμε μια δουλειά με στόχο την απλοποίηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μένα, ταυτόχρονα όμως ότι με τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ούτε τις βασικές αρχές ούτε και τις, τους στόχους της πολιτικής της συνοχής, μας οδηγεί στο να υπογραμμίσουμε τον στρατηγικό χαρακτήρα της πολιτικής συνοχής όπως ορίζει το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, βλέπουμε την συνάφεια μεταξύ της έκθεσης για την ε, πολιτική της συνοχής και τις μακροοικονομικές προοπτικές. Ταυτόχρονα όμω θέλω και να υπογραμμίσω ότι αυτό δεν μπορεί ποτέ να θέσει ένα αμφιβόλο την ε, εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής. Θα ήταν εσφαλμένο λοιπόν και ανέφικτο το να επαναδιατυπωθεί ο όρος ε, μακροοικονομικός. Επίσης η μακροχρηματοδότηση βεβαίως έχει σημασία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να, βγούμε από την, να ξεφύγουμε από την παγίδα που μερικές φορές κινδυνεύουμε να πούμε της παγίδας της συνοχής όταν έχουμε να κάνουμε πολιτικές όχι συμπληρωματικές αυτών των κρατών μελών στη συνεργασία τους, αλλά ε, που ουσιαστικά επαναφέρουν την εθνική διάσταση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη χρήση πόρων, μέσων χρηματοδότησης δηλαδή, και άρα έχουμε να κάνουμε με ένα ε, σημείο στο οποίο πρέπει να συλλογιστούμε με όρους λιγότερο ιδεολογικούς και περισσότερο ρεαλιστικούς. Ε, δηλαδή να κοιτάξουμε την αλήθεια και την πραγματικότητα κατά πρόσωπο. Με αυτέ τι δύο προκαταρκτικέ δηλώσει, που νομίζω καταγράφουν και τη συζήτηση που έχουμε κάνει μεταξύ μα, θα ήθελα να σα επιστήσω την προσοχή σε τρία ζητήματα πάνω απ' όλα, στα οποία, τα οποία με απασχόλησαν περισσότερο κατά την κατάρτιση των τροπολογιών. καταρχά η θεματολογία, η επιλογή της θεματολογίας. Και πολύ σύντομα, εδώ επαναφέρουμε το ζήτημα της θεματικής συγκέντρωσης, σε επίπεδο περιφερειακό και πάλι. Ε, η δική μου γνώμη τουλάχιστον είναι ότι είμαι κατά της εθνικού τύπου ή σε εθνικό επίπεδο συγκέντρωσης της θεματολογίας. Έτσι λοιπόν για τα θέματα, για τη θεματολογία προτείνουμε όχι να συμπληρώσουμε ή να διατυπώσουμε με λεπτομερείς όρους τα θέματα, αλλά να τα περιγράψουμε σε όρους γενικούς με μια μεγάλη πρόκληση που είναι το, η πράσινη Ευρώπη στο 30%, κύρια μεγάλη πρόκληση και μετά την άλλη μεγάλη πρόκληση μεταξύ των πέντε προτεραιοτήτων που είναι η μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτή προτείνουμε εμείς και θέλουμε ένα πεδίο εργασίας για τα ε, κράτη σε εθνικό επίπεδο δηλαδή, και ως προς τη συλλογή των δικτών που θα προέρχονται από τις περιφέρειες. Με καλύτερη ευελιξία λοιπόν για τη δεύτερη αυτή προτεραιότητα. Ξέρετε εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει ορίσει ως δεύτερο μεγάλο στόχο την καινοτομία, την έρευνα, την καινοτομία και δεν πρέπει να τον υποτιμούμε τον στόχο αυτόν. Ωστόσο, δίνεται η εντύπωση πως έχει παρουσιαστεί αυτή η πρόταση ότι ο στόχος είναι να υπηρετήσουν περισσότερο τις επιχειρήσεις τον επιχειρησιακό ε, σχεδιασμό και όχι τον εδαφικό, που δεν είναι όμως αυτό το μέλημα των κρατών και των περιφερειών. Ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα, στο οποίο θα σας παρακαλέσω και να συμβάλλετε και να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή, είναι η τεχνική υποστήριξη. Ναι, που όμως πρέπει να ενισχυθεί ιδιαίτερα με το τρόπο, με, τη θεματολογία του πώς αυτή η τεχνική υποστήριξη μπορεί να υπηρετήσει το στόχο, να ενισχύσει το διοικητικό δυναμικό. Πώς δηλαδή μπορούμε και μέσω των πόρων που διαθέτουμε στις περιφέρειες να βοηθήσουμε στη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα στο οποίο και ευαισθησία μεγάλη υπάρχει και ενδιαφέρον και αυτό αφορά όχι μόνο την Νότια Ευρώπη αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχει η βούληση για μια δημόσια διοίκηση που θα έχει χτιστεί έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγάλες προκλήσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τα κράτη και οι περιφέρειες δηλαδή πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Και να μην εκτίθεται πάντα σε μια τεχνική υποστήριξη εξωτερική της διάστασης του κράτους ή της περιφέρειας για τα ευρωπαϊκά θέματα, για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Ένα άλλο τρίτο θέμα, σημαντικό και μεγάλο, σε σχέση με την εδαφική συνοχή και έχω συλλέξει εδώ προτάσεις και ιδέες και των τοπικών περιφερειακών φορέων, είναι η ε, ιδιαίτερη έμφαση στην διάσταση την αστική των αστικών κέντρων. Κυρίως λοιπόν τα αστικά κέντρα έχουν προτείνει όχι ένα 6% που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ένα 10% των πόρων να αφιερωθεί στις, ε, στα αστικά κέντρα. Βεβαίως, με την επιφύλαξη ότι αυτό το 10% δεν θα περιορίζεται αυστηρά στο ακρικό κέντρο, αλλά θα απευθύνεται και στα, στις απομακρυσμένες περιφέρειες, τις ορεινές, τις μειονεκτικές, εκεί που έχουμε ε, απερίμωση, εκεί που έχουμε απώλεια πληθυσμού, εκεί που εντοπίζεται σε μεγάλο βαθμό και ε, τα, εντοπίζονται τα αίτια της, ε, στα, λόγω των αιτίων της κρίσης η αδυναμία της διαφύλαξης ενός κοινωνικού ιστού και συνοχής. Αυτό είναι το τρίτο μεγάλο θέμα λοιπόν, το οποίο προσπαθούμε να αναπτύξουμε μέσα από τις 72 τροπολογίες 44 που αφορούν το κείμενο. Για το Ταμείο Συνοχής, το την υπαριθμό 32 δηλαδή η τροπολογία, προτείνουμε την κατάργηση του άρθρου 5 της δεύτερης παραγράφου με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 10 δισεκατομμύρια ευρώ για το μηχανισμό προκειμένου να διατηρηθούν τα ποσά αυτά στο Ταμείο Συνοχής. Να παραμένουν τα ποσά λοιπόν αυτά ως ποσά συνοχής και αυτές εν ολίγης ήταν οι δικές μου ιδέες και σκέψεις σε σχέση με, ε, που εκφράζονται μέσα από τις 72 τροπολογίες μου και βέβαια είμαι στη θέση για να ακούσω τις προτάσεις και ιδέες των συναδέλφων λαμβανομένου υπόψη ότι έχουμε αρκετά σύντομα περιθώρια για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας με τα ε, τελικά σχόλια και αποφάσεις και εδώ στην Επιτροπή αλλά και στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστούμε κύριε Κοτσούλα. Τώρα το λόγο έχουν σκιώδεις συγητές και θα ακολουθήσουν άλλα μέλη της Επιτροπής ε, Ρέτζη. Και βέβαια έχουμε και τον προσκεκλημένο μας από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τον κύριο Βαρδακαστάνη. Ελπίζω να το πρόφερα καλά. Ναι, σας βλέπω. Είστε εκεί πίσω. Και μετά θα μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς όμως η εκπρόσωποι των κομμάτων. Κύριο Φαλκάλ Σελσίσο πρώτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την αρχική πρότασή του που είναι μια πολύ καλή βάση την οποία θα ε, αξιοποιήσουμε για να εμπλουτίσουμε το κείμενο της Κομισιόν. Όπως ε, είπαμε και στην ανταλλαγή απόψεων ε, Στόχος είναι να αναλύσουμε τα άρθρα 2 και 3 αναλυτικά, τα άρθρα που αφορούν δηλαδή τους στόχους αφενός και τη θεματική κέντρωση Θεωρώ ότι καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία ώστε οι τοπικές περιφερειακές αρχές κυρίως να μπορούν να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα ευελιξίας κατά τη διαχείριση των κονδυλίων. Τροπολογίες του εισηγητού προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουν. Είναι σημαντικό όμως από την άλλη πλευρά να μην αλλοιώσουμε την ε, θεματική συγκέντρωση ε, ούτε και την έμφαση που δίνει στα θέματα της ε, καινοτομίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ό,τι αφορά ε, τα στρες. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, δούμε ποια είναι τα κριτήρια που ορίζει το άρθρο 3 ε, σε ό,τι αφορά την εκ των προτέρων ρησιμότητα που τροποποιεί τώρα ο Σε ό,τι αφορά το γενικό πλαίσιο, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα σοβαρέ πτυχέ που δημιουργούν προβλήματα στι περιφέρειε. Παίρνουμε χάρη γέρανση του πληθυσμού ή απερίμωση που κινδυνεύουν να αφήσουν ε, άδειε, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, κάποιες περιφέρειες. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ πρέπει και μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σημερινή Ευρώπη. Καταλαβαίνω ε, και αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε ό,τι αφορά τη διαχείριση καταστροφών. Σεισμοί, ξηρασίες, πλημμύρες πρέπει να περιληφθούν ε, σε ενδεχόμενες τέτοιες ε, αιτίε ο ε, τυφώνας Λέσλι, μεγάλες πλημμύρες στις Βαλαρίδες για παράδειγμα. Είναι σαφή, ξεκάθαρα παραδείγματα το ότι πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στις περιοχές αυτές αλλά και στους πληγέντες από τέτοιες ε, διεξοκαιρικέ συνθήκες. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Ε, πρέπει να εφαρμόσουμε στην πράξη την αρχή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, να βοηθήσουμε ε, τους πληθυσμούς που τους ε, χτυπά με μεγάλη δύναμη η φύση και τους γείτονε. θα πρέπει η βοήθεια να διοχετεύεται με αποτελεσματικό τρόπο και να φτάνει το στομότερο δυνατόν στους ανθρώπους που τη χρειάζονται. Επίσης, νομίζω ότι όλα τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με το άρθρο 6 θα πρέπει να είναι τα πλέον κατάλληλα. Το λέει και ο εισηγητής άλλωστε. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των αποβλήτων, για παράδειγμα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ένα μοντέλο βιώσιμης κυκλικής οικονομίας, ολοκληρώνοντας. Καλό θα ήταν και ελπίζω να το λάβει υπόψη ο εισηγητή, να περιφθούν περισσότερε πρωτοβουλίε στο πλαίσιο τη αστική πρωτοβουλία ε, ε, και σε ό,τι αφορά τη διάθεση πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Άρθρο 9. Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνω εδώ την παρέμβασή μου, αλλά πρέπει να αποχωρήσω λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Δυστυχώ το πρόγραμμά μου δεν μου επιτρέπει, παρότι θα το ήθελα πάρα πολύ, να παραμείνω εδώ. Πρέπει μόνο να αποχωρήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα μπορέσετε να συνεργαστείτε με τον εισηγητή βέβαια, αφού είσαστε σκιώδης εισηγητής. Ο κύριος Πίτο έχει τώρα το λόγο. Σκιώδης εκ μέρους του ECR. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ξεκινώντας να αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο νομίζω προκύπτει κατόπιν ε, του τελευταίου γύρου συνομιλιών που είχαμε και ε, έχει να κάνει και με πολλά από τα ζητήματα που μας απασχόλησαν και ιδιαίτερα επιτρέπει να εξασφαλίσουμε ένα βήμα πρόοδου. Στα όσα είπε προκατακτικά ο εισηγητής μας, νομίζω ότι έχουμε και τα κύρια τις κυρίες απαντήσεις στα ζητήματα που μας απασχολούν. Θα ήθελα, χωρίς να επαναλαβώ αυτά που ήδη ακούστηκαν, να υπογραμμίσω κάποια ζητήματα αποφασιστικής σημασίας. Καταρχάς, Είναι πολύ σημαντικό να γίνει υπενθύμηση ότι δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολική συγκέντρωση. Καλύτερα ότι πρέπει να αποφευχθεί, να, να, να δεν πρέπει να λησμονηθούν ε, τελείωση λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Αυτό είναι μια επιλογή και σε σχέση με την οικονομική αλλά και σε σχέση με την τεχνική υποστήριξη γιατί πρόκειται για περιοχές οι οποίες έχουν μεγαλύτερη δυσκολία στην πρόσβαση και την κρίση αυτών των μέσων. Από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θετικό κρίνω και το ζήτημα των προτάσεων των σχετικών με την κλιματική αλλαγή για ολοκληρωμένη προσέγγιση και αποτροπή βέβαια των φυσικών καταστροφών θα πρέπει μεγάλη προσοχή να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις εργασίες μας, πιστεύω, πρώτον στο θέμα της στρατηγικής συγκέντρωσης πολιτικής συνοχής τα τελευταία χρόνια. Έχει αντιμετωπίσει ως ένας γενικό, έχει αντιμετωπίσει ως γενικό στόχο την πολυτομεακή πολιτική, τομε, πολυτομεακούς στόχους πολιτικής με συγκεκριμένες βέβαια προτάσεις και οράματα που όμως συν το χρόνο αποδείχθηκε ότι κατακαιρματίζει σε μεγάλο βαθμό την ορατότητα και την αποτελεσματικότητα. Έτσι λοιπόν η συγκεντρωτική θεώρηση πιστεύω η συγκέντρωση είναι ένας, ε, μια λύση που θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμίσουμε και να εδραιώσουμε. Μια δεύτερη παρατήρηση που ακούσαμε και από τον εισηγητή αλλά και από την προηγούμενη παρέμβαση ακούσαμε να επαναλαμβάνεται. Ε, θέμα καθοριστικό λοιπόν και για τις ε, καθαρά συμπληρωματικές ως προς την εθνική διάσταση οι πολιτικές και πρέπει να πούμε με απόλυτη σαφήνεια ότι υπάρχουν κράτη όπου οι πολιτικές της συνοχής έχουν ε, καταστεί μοναδική συγκεκριμένη πολιτική και μοναδικός πόρος ο οποίος απευθύνεται σε περιοχές με ιδιαίτερε δυσκολίες και αυτό δεν μπορεί να είναι παραδεκτό οπωσδήποτε. Θα πρέπει δηλαδή να εργαστούμε με συμπληρωματικέ πολιτικές και ταυτόχρονα θα έλεγα να απαιτήσουμε, να διεκδικήσουμε από τα κράτη-μέλη να επαναφέρουν ε, τον εστιασμό και τη στόχευση με τον ε, ιδιαίτερο στόχο και την απέτηση ε, της συνάφειας μεταξύ αυτής της πολιτικής συνοχής και του συμφώνου σταθερότητα, γιατί δεν μπορούμε να ε, λησμονούμε ότι υπάρχουν πόροι που θα πρέπει να δαπανώνται κατά τρόπο σωστό, δεν μπορούμε να εξουδετερώσουμε δηλαδή τον ε, συμπληρωματικό ε, χαρακτήρα και την υπηρεσία που προσφέρουν αυτοί οι πόροι και αυτά μέσα. Και τρίτον, ένα μεγάλο θέμα με χαρακτήρα πεστρό διαχειριστικό σε σχέση με τα προγράμματα και τον αριθμό των αρχών διαχείρισης. Προτάσεις για περιορισμό του αριθμού των αρχών διαχείρισης, παραδείγματι, μία αναταμείο για να μην έχουμε επικάλυψη μέσων τεχνικών που θα επιφέρουν συνέπειες διοικητικής επιβάρυνσης. Ε, μια τελευταία σκέψη που αφορά κυρίως ορισμένες χώρες Ας σταματήσουμε να μιλούμε με τίτλους και με επικεφαλίδες, αλλά ας στραφούμε πλέον στα συγκεκριμένα προγράμματα. Έχουμε δει ωραίες, ωραία αφηγήματα, χάρτες, ε, ε, γραφήματα που όμως εν τέλει δεν δίνουν τη δυνατότητα για μια συγκεκριμένη υλοποίηση, για συγκεκριμένα έργα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε πλέον τον τρόπο αυτή την πτυχή να την διευκρινίσουμε και κατά κάποιο τρόπο να την συνδέσουμε άρρηκτα με την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων. Εδώ λοιπόν έχουμε ανάγκη να εξασφαλίσουμε και να αξιοποιήσουμε μάλλον ένα θετικό κλίμα, αλλά και τη βούληση για συνεργασία σε όρους αγαστούς, για περισσότερη ε, ορατότητα και αποτελεσματικότητα πάνω απ' όλα της πολιτικής μας και πρέπει να βρούμε μέτρα ε, μέσα κατάλληλα για την υλοποίηση. Αυτόν άλλο στον δρόμο έχει χαράξει και ο εισηγητής. Υπάρχει αυτή η διαρκής αντιπαράθεση με την ιδέα της υλοποίησης. Είμαι βέβαιος ότι η έκθεση του θα οδηγήσει πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ είμαι η επόμενη σκιώδης εκ μέρους της Άλντε, οπότε επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω και τις πρώτες μου σκέψεις μετά την παρουσίαση της έκθεσης. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κύριο Κουτσουλίνο, τον εισηγητή, για την προετοιμασία του νομοθετικού αυτού κειμένου. Τα αρχικά μου σχόλια τώρα. Πρώτον, στηρίζω τον εισηγητή που λέει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα, συνεργειακές δράσεις και ευελιξία. Και κυρίως με το Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ πρέπει να συμπληρώνεται η εδαφική προσέγγιση με την προσέγγιση για μια περισσότερο κοινωνική Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Τώρα, όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων, από 25% σε 30% αυτή θα είναι η τροπολογία και τη στηρίζω απόλυτα. Στηρίζω δηλαδή τον εισηγητή σε αυτό. Στηρίζω και τον εισηγητή σε μια άλλη βασική τροπολογία να συμπεριληφθούν μέτρα για μηδενικές εκπομπές, προστασία ε, του φυσικού περιβάλλοντος, τον τουρισμό, γιατί πιστεύω ότι όντως τις εδαφικές, κοινωνικές και άλλες ιδιαιτερότητες των δικαιούχων πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας να υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο θεματική συγκέντρωση για την περιφερειακή κατηγορία, που να μην αλλάζει με πάνω από 10% όπως προτείνει ο εισηγητής. Τον στηρίζω επίσης για την αστική ανάπτυξη και την αύξηση 10% σε σχέση με το συνολικό ποσό. Και επίσης να ενισχυθεί η θεσμική και διοικητική ικανότητα ώστε οι δημόσιες αρχές και τοπικές αρχές να είναι πιο αποτελεσματικές κάθε φορά που χρησιμοποιούν κονδύλια του ΕΤΠΑ ή του Ταμείου Συνοχής. Στις διαπραγματεύσεις με τους συζητητές τα συζητάμε πάντα αυτά, γιατί για την ευελιξία συμφωνώ με το 5% σε θελοντική βάση μεταφορά στο ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής από το Invest EU ή άλλα μέσα. Και επίσης η σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πιστεύω ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις βάσει των συστάσεων που γίνονται, γιατί έτσι δημιουργείται μια μόχλευση της στήριξης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θέλω επίσης να στηρίξω και τη μεταφορά 10 εκατομμυρίων στην διευκόλυνση Connecting Europe για την περίοδο 2014-2020 και να λάβουμε υπόψη μας και τα προγράμματα που υπάρχουν για τις μεταφορές και για την προσβασιμότητα. Επίσης ευχαριστώ και για την εισαγωγή της καινοτομίας, που είναι μια εγκάρσια αρχή και σωστά πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα αριθμό 1. Δεν συμφωνώ με τη διαγραφή της πρότασης της Επιτροπής δυνατότητας δυνατότητας χρήσης των κονδυλίων σε rolling stocks, στις μεταφορές. Για καλύτερη κινητικότητα και μεταφορές με πολλά μέσα, πολυτροπικές μεταφορές. Προσβλέπω πάντως τη συνεργασία με τον εισηγητή και θα υποβάλω τις τροπολογίες μου. Προσβλέπω επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η απόψή μου ω και εισηγήτρια. Μαρτίνα Μισελ είναι η επόμενη, αλλά δεν είναι εδώ. Ο κύριος Σκέρλε τώρα που είναι σκιώδης εισηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για την παρουσίαση της έκθεσής του. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα αποτελέσει μια στέρεα βάση για παρετέρω συζητήσει και τροποποίησεις. Θα υποβάλω και εγώ τροπολογίες για να βελτιωθεί η έκθεση. Γενικά μιλώντας, πάντως πιστεύουμε ότι τοποθετείται σωστά ο εισηγητής και γι' αυτό πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε στα διάφορα σημεία της έκθεσης στηρίζουμε του να επιστρέψει το έτφα στις κοινέ διατάξεις. Το ίδιο και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για την ταξινόμηση πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει επιπλέον στήριξη. Η επίτευξη του στόχου 2 είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Για το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή πρέπει να αποτελούν την προτερότητά μας. Μόνο με βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να αναπτυχθεί παρετέρω η Ευρώπη. Και κάτι άλλο που εμένα με καίει πολύ είναι η κυκλική οικονομία. Και πιστεύω ότι έχει θέση και εδώ σε αυτή την έκθεση. Η πρόταση της Επιτροπής για την διαχείριση αποβλήτων είναι καλό. Είναι η καλύτερη πηγή χρηματοδότησης το ΕΤΠΑ και η συνοχή για πολλές ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να πετύχουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ηγηθεί όσον αφορά το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Έχουμε να πετύχουμε πάρα πολλούς στόχους μέχρι το 2027 και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς, τα αναπτυξιακά μας σχέδια και προγράμματα πρέπει να τους λαμβάνουν υπόψη. Αυτό το νομιθετικό πακέτο για την διαχείριση αποβλήτων και η Συμφωνία των Παρισίων πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις ρυθμίσεις μας. Η κυκλική οικονομία επίσης αναφέρεται στο δεύτερο στόχο, αλλά θα πρέπει να εισαχθεί και στον πρώτο στόχο. Γιατί πρέπει να αναγνωριστούν στην Ευρώπη τα πλονεκτήματα της κυκλικής οικονομίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, επιχειρήσεων πρέπει να λειτουργούμε βάσει των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Οι νομοθέτες πρέπει να στείλουν ένα σαφές μήνυμα επίσης όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής. Τα κονδύλια πρέπει να πιάνουν τόπο, να στηρίζουν τους περιβαλλοντικούς στόχους ακόμα και αν δεν αυξάνεται έτσι η ανταγωνιστικότητα ή δεν υπάρχουν οικονομικά ωφέλη ε, βραχυπρόθεσμα. Όμως τα κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη μπορεί να αποδειχθούν τεράστια αργότερα, μακροπρόθεσμα. Προσβλέπουμε και εμείς σε συνεργασία με τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές για αυτό το θέμα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Ανταμάτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ τον συνάδελφο. Η πρόταση του νέου κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής ε, πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη το, το εξή δεδομένο ότι σε, για διάφορου λόγου το Ταμείο Συνοχή, ε, πολλά κράτη-μέλη ε, καλύπτουν το 50% των δημόσιων ή αντιστοιχούν στο 50% των δημοσίων ταπανών. Βεβαίω, και με αυτή τη θετική τόνα, με αυτό το θετικό τόνο, με αυτό το θετικό κλίμα μπορεί να ξεκινάμε, αλλά ταυτόχρονα ε, καθίσταται κάπως πιο αρνητικό το κλίμα, το βλέπουμε τι προτάσεις διατυπώνονται. Εδώ έχουμε κάποιες στρατηγικές λοιπόν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εφίους ε, Συνεργασίες που υποκαθιστούν τις επενδύσεις και, τα, και υποτίθεται ότι φέρνουν και προσθεμένη αξία του, τα πλεονεκτήματα όμως θα τα δούνε μόνο οι πλέον ανεπτυγμένες περιοχές. Πρέπει να γίνει προσπάθεια λοιπόν για καλύτερα αποτελέσματα σε όλες τις περιφέρειες. Είναι θετικό το λεγόμενο earmarking του 6% για το ΕΤΠΑ, για την ανάπτυξη των αστικών κέντρων, αλλά εγώ θα ήθελα να αυξηθεί το ποσοστό αυτό. Είναι πολλές οι προκλήσεις ενταξύ των μεταναστών, κοινωνική ενσωμάτωση που μπορούν ε, να καλυφθούν ε, και να καλύψουν τις ανάγκες των αστικών κέντρων. Ε, ίσως θα πρέπει να προβλέψει ένα ειδικό μέτρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τα αστικά κέντρα που θα κάλυπτε τις ανάγκες των πολιτών των αστικών κέντρων ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ενεργειακή μετάβαση, κινητικότητα και πολλά άλλα. Ε, οι στρατηγικές που προβλέπονται ε, στον προγραμματισμό 2014-2020 και είναι θετικές μεταφράζονται σε ολοκληρωμένα περιφερειακά προγράμματα στις περιφέρειες ε, με προγράμματα συμμετοχικά οι φορείς, οικονομικοί, κοινωνικοί φορείς διαφόρων επιπέδων συμμετέχουν και συνεργάζονται με τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές και αυτή τους συμμετοχή έχει κέρια σημασία και για τον προγραμματισμό αλλά και για την, ε, στην πράξη υλοποίηση. Δηλαδή και σχεδιασμός και εφαρμογή. Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι η αναφορά σε μη χρηματοδοτούμενα έργα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, αυτά δηλαδή τα οποία θεωρεί ότι δεν συνάδουν με την ε, συνοχή. Καπνοβιομηχανία, χωματερές, πυρηνικά εργοστάσια. Σημαντικό επίσης είναι να υπογραμμιστεί το Ταμείο Συλλογής πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι και απαραίτητο για τα άτομα με αναπηρία από τη λεγόμενη institutional care ιδρυματική δηλαδή υποστήριξη, στην υποστήριξη από την οικογένεια ή στον εγγύς κοινωνικό ιστό για τα άτομα με αναπηρία. Το βλέπουμε στην πρόταση της Επιτροπής, θα ήθελα όμως πιο πολλές ε, διευκρινήσεις, τις οποίες θα υποβάλω μέσω των τροπολογιών μου. Τώρα όμως τις επικρίσεις, αφού είδαμε τα θετικά. η θεματολογία και η στόχευση σε εθνικό επίπεδο, που επεσήμανε και ο συντάκτης μας θα είναι πολύ δύσκολο στην πράξη να υλοποιηθεί ε, αυτός ο στόχος και η μεγαλύτερη ευελιξία που προτείνει και ο κύριος Κοτσολίνο με την κατανομή σε όρους περιφερειακούς είναι πολύ πιο λογική. Και έτσι και εμείς θα κάνουμε τις δικές μας τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Με ανησυχεί επίσης το θέμα της συνέργειας που αναφέρεται ως όρος ε, για τα κονδύλια του ΕΤΠΑ. Βεβαίως οι αγαστές συνεργίες, το ορίζον, το excellence, η έννοια της αριστείας δηλαδή, είναι πολύ σημαντικές έννοιες. Αλλά Μα ανησυχεί το γεγονό ότι ένα 5% των ταμείων συνοχή θα μπορούν τα κράτη-μέλη να το μεταφέρουν στο Invest Europe, το λεγόμενο την τρίτη εκδοχή του πακέτου Juncker. Έτσι λοιπόν, αν δεν υπάρξει μία συγκεκριμένη στόχευση για περιφέρεια συγκεκριμένη των ποσών αυτών ε, κινδυνεύουν να χαστούν τα κονδύλια κάπου αλλού. Η μακροοικονομική αιρεσιμότητα δεν μας βρίσκει σύμφωνος και πιστεύω ότι πρέπει ε, αντί για το δημόσιο έλλειμμα τα κονδύλια να χρηματοδοτούν τις ανάγκες των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και οι τροπολογίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποστινάρου, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ μας. Ήμουνα νωρίτερα εγώ εισηγητής για το Ταμείο Συνοχής, οπότε προσφέρθηκα να βοηθήσω τον Ανδρέα και να συνεργαστούμε για το σχεδιασμό του νέου τμήματος συνοχής στην έκθεση. Και καταφέραμε, πιστεύω, να πετύχουμε ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα. Και θα αναφερθώ σε ένα ζήτημα πρώτα απ' όλα που μας απασχολεί όλους. Τροπολογία 5 όπου συζητάμε την ικανότητα και τη δυνατότητα των χωρών μελών να αντιμετωπίζουν από κοινού φυσικές καταστροφές και από κοινού να προσφέρουν διαχείριση στην περίοδο μετά την κρίση ή μετά την καταστροφή. Η Ρουμανία οργάνωσε τη μεγαλύτερη άσκηση μετά από σεισμό του 2018. Κινητοποιήθηκαν άνθρωποι από το Υπουργείο Εσωτερικών, Άμυνας, γιατροί. Ο μελητής μιλάει εκτός μικροφώνου και τον ακούμε δύσκολα οι Ηνωμένε Πολιτείε το κάνουν. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή κινητοποίηση, πρέπει να πω. Και ο Επίτροπος Τηλιανίδης ήρθε στο Βουκαρέστι και ήταν η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τέτοια άσκηση που μας επέτρεψε να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, πρώτον για να αποφεύγουμε καταστροφές και δεύτερον για να αντιμετωπίζουμε καταστροφές, βελτιώνοντας μάλιστα ε, κανόνες και ρυθμίσεις ώστε να μπορούμε πιο γρήγορα να προσφέρουμε βοήθεια και να μετοπίσουμε την καταστροφή. Και θα τελειώσω με το συμπέρασμα του Επιτρόπου Στυλιανίδη. Δεν υπάρχει δυνατότητα από μόνη της μία χώρα μέλος να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και ικανοποιητικά σε καταστροφή μεγάλης κλίμακας. Από κοινού όμως ως Ένωση μπορούμε. Τώρα, για άλλα ζητήματα. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα του προπολογισμού πρώτα απ' όλα. Το Ταμείο Συνοχής έχουν γίνει όμως περικοπές και γι' αυτό επιμένουμε να βρεθεί κάποια διευθέτηση στο μέλλον, στο μελλοντικό δηλαδή πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε αν μη τι άλλο να πετύχουμε το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης που έτσι κι είναι χαμηλό. Η μεταφορά τώρα των 10 εκατομμυρίων στη διευκόλυνση για την Ευρώπη. Χαίρομαι για την απόφαση που πήραν και οι συγητές και οι συντονιστές κατά της μεταφοράς αυτής. Για ποιο λόγο. Γιατί όσο έχουμε περικοπές και ζητάμε μεταφορά 30% του Ταμείου Συνοχής στην κεντρική διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για μένα και για μας αυτό είναι κάτι αδύνατον. Αλλά πρέπει να υπάρχουν ευέλικτες λύσεις, να τις εντοπίσουμε για να δούμε πόσο μπορούμε να μεταφέρουμε έτσι, ναι. Αλλά μόνο εάν έχουμε μια καλύτερη απάντηση από την Επιτροπή από ό,τι έχουμε τώρα. Κάποια άλλα σημεία όπου συνεργαστήκαμε με τον Αντρέα, ενίσχυση της διοικητικής και θεσμικής ικανότητας. Και εδώ ευχαριστώ τη στήριξη όλων των συναδέρφων. Επίσης, ενίσχυση της ιδέας ότι κάθε χώρα συνοχής θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει πόσο θα επενδύσει σε προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον και πόσα σε ευρωπαϊκά δίκτυα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε χώρας. Γι' αυτό μιλάμε για ευελιξία και ελπίζω οι συνάδελφοι να στηρίξουν την πρότασή μας αυτή. Τι αποκλείεται τώρα. Επιμένω και σας παρακαλώ προσέξτε μου στο θέμα της θέρμανσης, άνθρακας λοιπά Είναι στοιχεία πολύ σημαντικά για πολλές χώρες. Όμως, αναφέρομαι κυρίως στο γεγονός ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την επιλεξιμότητα ώστε να βελτιωθούν περιφερειακά συστήματα θέρμανσης κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα προβληματικό στις χώρες Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Και ιδίω τώρα μετά, τις, ε, μετά την κλιματική αλλαγή είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πώς θα περάσουμε το χειμώνα. Μερικές φορές οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές. Γι' αυτό και επιμένουμε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα επιλεξιμότητας προγραμμάτων που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα και κυρίως στο φυσικό αέριο. Και γιατί φυσικό αέριο. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι η πιο οικολογικά συμβατή ε, πηγή και ίσως γι' αυτό έπρεπε να έχει αναπτυχθεί το Nord Stream. Αλλά μην ξεχνάμε συνάδελφοι ότι χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την ενεργειακή μετάβαση προς ε, πιο φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή ενέργειας. Και ένα στοιχείο που έχω κατά νου είναι η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας με το district heating, με την ε, μόνωση των κτίριων. ...36 με 40% μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να έχουμε πιο καθαρό περιβάλλον. Αυτό δείχνουν διάφορες μελέτες. Η δικιά μου τροπολογία έχει να κάνει με την ίδια φιλοσοφία όπως και την προηγούμενη φορά. Σας είπα. Και δεν επηρεάζει το σύστημα εμπορίας εκπομπών, το ETS. Να επιτραπεί λοιπόν η καύση και να αναφερόμαστε μόνο στο φυσικό αέριο. Άλλα στοιχεία σε σχέση με αυτά που αποκλείονται. Ευχαριστώ την Πρόεδρο για τα σχόλιά της. Συμφωνώ. Και η δικιά μου τροπολογία προστίθεται σε αυτή την ιδέα. Γιατί υπάρχουν πολλές χώρες μέλη που προσπαθούν να βελτιώσουν, να βελτιώσουν τα, τις μεταφορές τους και χωρίς τη στήριξη των Rolling Stocks αυτό είναι δύσκολο. Το τροχαίο υλικό δηλαδή. Πρέπει να στηριχτεί και η τροπολογία του εισηγητή από αυτού. Τέλος. Ευχαριστώ και για τη θεματική συγκέντρωση σε περιφερειακό επίπεδο και όχι σε επίπεδο χώρας μέλους. Γιατί αντικείμενο της περιφερειακής πολιτικής είναι οι περιφέρειες, όχι χώρες. Γι' αυτό να γίνεται μνήα στις περιφέρειες και να υπάρχει παραπάνω ευελιξία στις περιφέρειες να μπορούν να επιλέξουν θεματικά και να επικεντρώσουν εκεί τους πόρους τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Συμφωνώ βέβαια ότι πρέπει να υπάρχει και ένα επίπεδο κριτηρίων. Αλλά να υπάρχει σαφώς βαθμός ευελιξίας για τις περιφέρειες, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρο. Κύριος Μοσκούρ, παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου. Sorry. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στη δική σας ε, την παρέμβαση μιλήσατε για τη σημασία του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής για την ανάπτυξη των ε, εδαφών ε, και ιδίως των νησιωτικών περιοχών. Η έκθεση μου φαίνεται λοιπόν προς το σημείο αυτό πολύ σημαντική και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ποιοτική δουλειά που έχει κάνει. Είναι πραγματικά πολύ ε, καλή έκθεση γιατί αναλύει, ε, δίνει ευελιξία και νομίζω τελικά ε, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Στηρίζω και τις προτάσεις για τον επαναπροσδιορισμό τη θεματική συγκέντρωση σε περιφερειακό επίπεδο, όπως υπόθηκε. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προωθούμε την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή εγγύς των περιφερειών. Είμαστε κατά της υπερβολικής ε, συγκέντρωσης βέβαια. Θέλω επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την πρόταση του εισηγητή σε ό,τι αφορά τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Τουλάχιστον 30% θα χρησιμοποιήσουν, τη χρηματοδότηση δηλαδή, για να στηρίξουν επιχειρήσεις ε, υπέρ μιας πράσινης Ευρώπης, ώστε ιδίως οι εξόχω απόκεντρε περιφέρειες που είναι ευάλωτε ε, σε φυσικές καταστροφές ε, θα μπορέσουν να ενισχύσουν την αντοχή τους και τη δυνατότητα πρόληψης αλλά και διαχείρισης κινδύνων. Βέβαια, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, θα καταθέσω και εγώ τροπολογίες, διότι νομίζω ότι το κριτήριο ταξινόμησης των περιφερειών στο άρθρο 3 νομίζω ότι θα έπρεπε να ανταποκρίνεται πιο καλά στις διαφορετικές πραγματικότητες ε, αν λαμβάνονταν υπόψη το ΑΕΠ και η αγοραστική δύναμη ταυτόχρονα. Επίσης, θέλω να καταθέσω τροπολογία να δούμε ποιοι είναι θετικοί αντίκτυποι, συγκεκριμένοι επιπτώσεις. Ε. Έχουμε το άρθρο 11 κανονισμού αυτού που νομίζω ότι θα πρέπει να επιτρέπει τη χρηματοδότηση μηχανισμών εδαφικής συνέχειας. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε να προωθήσουμε την κινητικότητα των Ευρωπαίων που ζουν σε υπερπόντια εδάφη και να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, κύριε Μπόκοβιτς, σας παρακαλώ. Πρόεδρε, εδώ έχουμε να κάνουμε μια έκθεση πολύ σημαντική. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Είναι πολύ καλά προετοιμασμένο το σχέδιο. Και βλέπουμε αναγυγνώμης κοντά στο πως η περιφερειακή πολιτική ανάπτυξη της Πέθρου ε, βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση υπογραμμίζει πολλά θετικά και βελτιώνει πολύ το κείμενο. Θα συμφωνήσουμε τόσο υπόθηκαν και όσα έχουμε κάνει και με άλλες εκθέσει. Θα πρέπει να αγωνιστούμε, να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε το επίπεδο χρηματοδότησης. Ε, ο... Για τον κανονισμό τώρα κοινών ε, διαδικασιών. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε μια λύση συμβιβαστική, ε, φερρυπίν, ε, ότι Ε, υπάρχει και η εδαφική διάσταση πέραν της διάστασης της περιοχής της Υπέθρου ή κάτι αντίστοιχο. Μπορούμε νομίζω να βρούμε μια λύση για μια καλή κοινή διαχείριση. Όσον αφορά τις προτάσεις του εισηγητή. Η κλιματική διάσταση, η διάσταση της κυκλικής οικονομίας, ε, και άλλες, νομίζω είναι ξεκάθαρα ορατές μέσα στην πρόταση. Στα αστικά κέντρα βλέπουμε ότι χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη, γιατί αυτά είναι και ο κινητήριος ε, ε, μοχλός της ανάπτυξης. Ιδιαίτερη μνήα γίνεται και στις απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές αλλά και τις περιοχές της Υπέθρου και τις ορεινές περιοχές θα έπρεπε να αναφέρουμε. Άλλωστε το είχαμε περιλάβει και στο κείμενο του ψηφίσματος στο παρελθόν και πιστεύω θα πρέπει να βρούμε μια λύση γιατί εάν δούμε το, στη συνολική χρηματοδότηση η πολιτική της συνοχής, η περιφερειακή ανάπτυξη ε, έχουν πρόβλεψη μικρότερων κονδυλίων. Πολύ φοβούμαι ότι αυτό το κομμάτι του προϋπολογισμού δηλαδή θα ε, περικοπεί σημαντικά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επαγρυπνούμε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Άλλωστε είναι πολλοί αυτοί που εγκαταλείπουν την Ήπεθρο και μετακινούνται στα αστικά κέντρα ή εγκαταλείπουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες ε, περιοχές των κρατών μελών για να, μεταβούν, να κατασταθούν σε πιο ανεπτυγμένες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε τη χρηματοδότηση όπως την προβλέπει το σχέδιο του προπολογισμού. Αυτό θα το επιδιώξω και εγώ με τις τροπολογίες μου φυσικά. Ε, για τα ευφύ χωριά, παραδείγματι, χρειαζόμαστε σαφή οράματα για τις περιοχές αυτές. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω και κάτι ακόμα. Ε, στην ανοικοδόμηση, αποκατάσταση, πρέπει να έχουμε την ενεργειακή διάσταση, αλλά και όταν μιλούμε για ε, σεισμούς και φυσικές καταστροφές, πρέπει να βελτιωθεί ο τρόπος ανέγερσης των κτηρίων, ώστε να είναι πιο ανθεκτικά στις σεισμικές δονήσεις. Θα το επιδιώξω αυτό και μέσω των τροπολογιών μου. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κάποιος άλλος από τους συναδέλφους της Επιτροπής μας, κύριε Φανίστηλ Ρόη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, ο οποίος νομίζω ότι πάρα πολύ καλά έχει συμπεριλάβει όλα όσα σκεφτόμαστε εμεν και δε. Την ευελιξία, τις επιλογές που πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους οι περιφέρειες, είναι κάτι που το θέλει και η Επιτροπή των Περιφερειών, το έχουν πει. Έχω μια ερώτηση. άρθρο 3 για τον προπολογισμό και στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περιμένω αντιδράση. Σε περιφερειακό επίπεδο μιλάμε για το κατακεφαλή ΑΕΠ, ενώ η Επιτροπή έχει επιλέξει την εθνική διάσταση, δηλαδή το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα. Δεν είναι μόνο θέμα όρων, ποιες ε, είναι οι επιπτώσεις της μία περίπτωσης και της άλλης περίπτωσης. Όσον αφορά τις περιφέρειες, αυτό θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας το εξηγήσει. Τι σημαίνει αυτό για τις περιφέρειες, για την κατανομή των πόρων. Έχει τόσο μεγάλη σημασία, θα μπορούσε να είναι ή το ένα ή το άλλο. Αδιακρίτως. Άκουσα τη συζήτηση και ένα σχόλιο έχω να κάνω. η οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Η γνώση είναι κάτι πολύ γενικό. Εμείς είμαστε πλούσιες περιφέρειες, λέμε ότι έχουμε γνώση, η Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα το είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ολόκληρη την Ευρώπη, για την Νότια Ιταλία, για, για όλους. Πρέπει να είναι ένα δημόσιο αγαθό αλλά τότε οι επιχειρήσεις πού βρίσκονται. η γνώση, άμα μοιράζεται για να παράγουμε νέα προϊόντα βασισμένη στη γνώση. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με τις επιχειρήσεις όμως, γιατί οι επιχειρήσεις τα ελοποιούν όλα αυτά. Να χρηματοδοτείται η εφαρμοσμένη γνώση και να υπάρξει δίκευση στις περιφέρειες. Δεν μπορεί κανείς να είναι καλό σε όλα άμα θέλεις να είσαι καλό σε όλα, χάνεις τη, το αντιγωνιστικό σου πλεονέκτημα σε σχέση με όταν ειδικεύεσαι σε ένα πράγμα. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό στους καιρούς που ζούμε. Ίσως είναι καλύτερα ο καθένας να επιλέγει το δικό του τομέα και να τον δουλεύει παραπάνω για να γίνει πιο καλός σε αυτό. Αυτά. Ε, εντάξει, για τις επιλογές των περιφερειών, ναι, συμφωνώ. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που πάντα συζητάμε εδώ. Να ενισχύσουμε και την πόλη και την Ήπεθρο. Να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός οι πόλεις να έχουν υπόψη τους και την περιφέρεια. Στο πρώτο άρθρο πρέπει να επανέλθουμε αν θέλουμε να δούμε ε, τους ορισμούς και τα περιπέθρου. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βαρδακαστάνης από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Παρακαλώ. Thank you, Madam President. First of all, I... Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να έρθουμε να σας παρουσιάσουμε το έργο μας για αυτό τον προτινόμενο κανονισμό για την περίοδο 2021-2027 σε ό,τι αφορά το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Η Επιτροπή μας πρώτα και πάνω απ' όλα επανεπιβεβαιώνει την ε, προσήλωσή της και την ε, πίστη της στην πολιτική συνοχής. Ταυτόχρονα εκφράζουμε και τη λύπη μας για τις περικοπές οι οποίες περιλαμβάνονται 10% συνολικά για την πολιτική συνοχή και 20% για το ΕΤΠΑΠ και 46% για το Ταμείο Συνοχής, για το ΣΥΕΦ. Και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να επαναφέρει τον προϋπολογισμό στα επίπεδα της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Συνολικά για την πολιτική συνοχή, αλλά και για ταμείο συνοχής και ΕΤΠΑ, ειδικότερα. Επίσης, στη γνωμοδότησή μας, υπογραμμίζουμε και τη διαφωνία μας με την αλλαγή στα ποσοστά σε χρηματοδότησης. Καλούμε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κριτήρια συγχρηματοδότησης να τα καταστήσει πιο ευέλικτα, έτσι ώστε η οικονομική, χρηματοπιστωτική κατάσταση των κρατών μελών αλλά και φυσικά και των περιφερειών να λαμβάνεται υπόψη. Και βεβαίως όλα αυτά σχετίζονται με τις μακροοικονομικές αιρεσιμότητες οι οποίες αποφασίζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και επιβάλλονται αν συνεχεία στις περιφέρειες. Κατά την άποψή μας πρέπει να είναι ευέλικτε ή αλλιώς να διαγραφούν. Πάντως, καλωσορίζουμε τις βελτιώσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στο μέτωπο της απλούστευσης και της ευελιξίας. Πάντως θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η απλούστευση και η ευελιξία δεν θα πρέπει να βάλουν κατά μέρος αξίες και αρχές που είναι στο, επίκεντρο και στην καρδιά του ευρωπαϊκού κεκτημένου, όπως είναι η ισότητα, η μη διακριτική μεταχείριση, προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Θα επανέλθω. Η Επιτροπή μας ε, καλωσορίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της βελτιώνει την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην επιμερισμένη διαχείριση και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων αυτής, αλλά και άλλων εμπλεκομένων φορέων, στη διαδικασία του προγραμματισμού, της εφαρμογής, αξιολόγησης και της Παρακολούθηση της χρήσης ε, των κονδυλίων. Ωστόσο, ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Συμπεριφοράς ε, για τις εταιρικέ σχέσεις θα πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστός σε, όλα τα επίπεδα. Εξού και με την πρόταση να θεωρηθεί αυτό ένας ευκολυτικός παράγοντας enabling condition. Επίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει οργανωμένος διάλογος με όλους τους ευλακωμένους φορείς ό,τι αφορά την πολιτική συνοχής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Φόρουμ Συνοχής, ώστε οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς να είναι πραγματικοί συμμετέχοντες και πρωταγωνιστές στη διαδικασία εφαρμογής στο πλαίσιο της νέας περίοδου προγραμματισμού. Η ΕΟΚΕ συστήνει να εξορθογήσει και να περιλάβει τη βιώσιμη ανάπτυξη, του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κομισιόν και στην πολιτική συνοχής αλλά και στον κανονισμό ΕΤΠΑ, Ταμείου Συνοχής. Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που δεσμεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει χωρίς επιφυλάξεις και ενδιασμούς ε, την ε, ατζέντα και το θεματολόγιο το σχετικό. Δεν έχουμε όμως δει μια στρατηγική για την εφαρμογή και συμπερίληψη αυτής της στρατηγικής 2030 σε όλες τις πολιτικές, εσωτερικές, εξωτερικές. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή τη σπουδαία ευκαιρία. για την πολιτική σχέση και στην προκειμένη περίπτωση για το Ταμείο Συνοχή ε, και το ΕΤΠΑΓΙΑ, τι αεροκατοικημένε περιοχέ, τα νησιά κτλ. Άκουσα τον εισηγητή και άλλου και συμφωνώ απολύτω μαζί του ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν τι περιοχέ αυτέ όπω ακριβώ και τι εξόχου απόκεντρε ε, περιοχέ. Πρόκειται για μεγάλο έλλειμμα στη πρόταση κανονισμού. Και θα θέλαμε η Επιτροπή σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι στην πρώτη γραμμή και να προωθήσουν ε, μια μείζων αλλαγή σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τα νησιά και τις αεροκατοικημένες περιοχές. Τώρα είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Δαφική Συνεργασία το Ιντερεκ να έχει περισσότερο προπολογισμό. και στη νέα περίοδο προγραμματισμού για να μπορεί να εκπληρώσει αποτελεσματικά την αποστολή της, τους στόχους της. Αν δεν δοθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την επίτευξη των στόχων, θα υπάρξει διαφορά και απόκληση μεταξύ έργων και λόγων. Κάτι που το βλέπουμε κάποιες φορές. Αυτό που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ΕΟΚΕ είναι να λάβει υπόψη και άλλους κοινωνικού δείκτες. Όχι μόνο το καθάριστο εισόδημα κατά την ε, συζήτηση της θεματικής συγκέντρωσης και την ταξινόμηση των περιφερειών. Το καθάριστο, το εθνικό καθάριστο εισόδημα δεν μπορεί να τα περιλάβει όλα και στηρίζουμε την αρχή θεματικής συγκέντρωσης. Καταλαβαίνουμε το συλλογισμό. του να λαμβάνεται η περιφέρεια ως βάση θεματικής συγκέντρωσης. Θέλω τώρα να αναφέρω κάποια άλλα σημεία συνδεδεμένα μεταξύ τους ε, στην ε, πρόταση βλέπουμε το 7 άρθρο για την ισότητα και την προσβασιμότητα με αναπηρία. Η λογική που έχει προβληθεί είναι ότι είναι σημαντικότερο να υπάρξει σε άλλα άρθρα, όπως είναι το άρθρο 67 για παράδειγμα του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, η πρόσβαση δηλαδή των ατόπων με αναπηρία δεν, εφάρμο, δεν ε, αναφέρεται. Θέλουμε να το κοιτάξετε αυτό, γιατί ο στόχος μας Μέσω του ΕΤΠΑ και της χρηματοδότησης και της χρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής πρέπει να αποσκοπούμε στη δημιουργία προσβάσιμων προσβάσιμων περιβάλλοντος. Πρέπει να λάβετε υπόψη το εξή. Έχουμε 80 εκατομμύρια Ευρωπαίους συμπολίτες μας με αναπηρία. Ο πληθυσμός γυράσκει. Όλο και περισσότερα εκατομμύρια συμπολίτες μας ε, παρουσιάζουν μειωμένη κινητικότητα. Ποτέ δεν θα πρέπει να αφήσουμε να μας ξεφύγει αυτή η πολύ, πολύ σημαντική ευκαιρία μέσω του ΕΤΠΑ, μέσω της πολιτικής συνοχής, για να έχουμε αυτά τα προσβάσιμα περιβάλλοντα, όπως τα είπα. και στο ψηφιακό τομέα, στις μεταφορές κτλ. Νομίζω η κυρία Νταμάτο ήταν αυτή η οποία ανέφερε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Έχει ήδη κυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το στηρίζουμε να συμπεριληφθεί και επίσης θα θέλαμε στο άρθρο για τις εξαιρέσεις όποια χρηματοδότηση παρέχεται για την δημιουργία, την αναμόρφωση ε, κλειστών χώρων ε, ιδρυμάτων ε, θα πρέπει να γίνει γιατί το κοινοβούλιο πρέπει να δείξει κόκκινη κάρτα εδώ. Αν πραγματικά θέλουμε να εφαρμοστεί ο κοινωνικός πυλώνας, πρέπει να δώσουμε βάση κοινωνικές υπηρεσίες για όλους όσους τις χρειάζονται στρέφομαι στις μακροοικονομικές αρισιμότητες. Μάλλον όχι, τα κάλυψα αυτά. Άρα ολοκληρώνω λέγοντας ότι συμφωνούμε με την αστική πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία Urban είναι μια πρωτοβουλία πολύ χρήσιμη και αν υπάρχει δυνατότητα αύξησης του ποσοστού χρηματοδότησης πρέπει να γίνει αυτό. Όμως, διαβάζοντας τον πρωτονόμο κανονισμό για το ΕΤΠΑ, το τέσσερα που αφορά τον ε, κοινωνικό πυλώνα είναι αδύναμο. Προτείνουμε λοιπόν η πρωτοβουλία κοινωνική βιωσιμότητα και προσβασιμότητα πρέπει να προωθηθεί με το 10%. Καταλαβαίνουμε ποιο είναι το επιχείρημα για το ΕΚΤΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, ότι θα στηρίξει αυτό την ε, υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όμω και το υπογραμμίζω, δεν μιλάμε μόνο για κατάρτιση, απασχόληση, υπηρεσίε κτλ. κτλ. Αν θέλουμε να έχουμε ένταξη, να μην έχουμε διακρίσεις και να έχουμε ισότητα, δεν φτάνουν αυτά. Χρειάζονται βιώσιμα περιβάλλοντα. Αηφορία, βιωσιμότητα, προσβασιμότητα, σημότη, συγγνώμη. Να μπορεί ο κόσμος να ζει με βάση προσωπικές του επιλογές. Πάντοτε είχαμε καλή συνεργασία με την ε, Επιτροπή σας και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που μας δώσετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την γνωμοδότηση μας η οποία θα εγκριθεί την επόμενη Τετάρτη επισήμω ε, στην Ολομέλεια της ΕΟΚΕ. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση των συναδέλφων της Επιτροπής μας. Έχουμε επίση και τον εισηγητή τη Επιτροπή των Περιφερειών προσκαλέστερα να επισημάνω. Δυστυχώ όμω δεν κατέστη δυνατό να συμμετάσχει σήμερα. Και θα προσπαθήσουμε βέβαια την συζήτηση να την αναπτύξουμε σε όσο δυνατόν πιο διαφανή τρόπο. Παρακαλώ τώρα τον κύριο Φανμπρέσκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβω το, το λόγο, βλέποντα ότι, επισημένοντα ότι η ομάδα τη Επιτροπή έχει εντωμεταξύ ενισχυθεί. Ναι, ναι, βεβαίω, γιατί τώρα μιλάμε για χρήματα. Καταρχά, σα ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Κοτσολίνο για την πολύ λεπτομερή δουλειά του στην έκθεση. Ε, πέντε παρατηρήσει αν μου επιτρέπετε. Καταρχάς θεματική συγκέντρωση και εδώ ε, πρέπει να ομολογήσω ότι μας ανησυχούν κάπως ε, οι αλλαγές που βλέπουμε ως προς τη, που προς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι η εφαρμογή σε περιφερειακό επίπεδο των ε, απαιτήσεων θεματικής συγκέντρωσης κατά την άποψή μας οδηγεί σε μια πιο περιοριστική σε σχέση με την εθνική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόταση, γιατί θα έχει σαν συνέπεια ε, να υποχρεωθεί κάθε περιφέρεια να περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Ενώ η δική μας πρόταση ε, επιτρέπει ευελιξία. Γιατί μια άλλη στο βαθμό που εξασφαλίζεται, με υπό την προπόθεση ότι εξασφαλίζεται εθνικός μέσος όρος. Ε, η προσθήκη μιας ε, ευελιξίας της τάξης του 10% δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζει τα προβλήματα άλλωστε. Αντιθέτως, ακόμη περισσότερο τα περιπλέκει, γιατί πρέπει να γίνεται η ανείχνευση ε, αυτής της κατάστασης και άρα είναι μεγαλύτερο ακόμη το δημοσιονομικό άχθος. Επιφυλακτικοί είμαστε επίσης ως προς την πρόταση της έκθεσης του σχεδίου έκθεση για την χρήση τουλάχιστον δύο ε, στόχων πολιτικής για, τους, για τις πιο ανεπτυγμένε ε, περιφέρειες. Εδώ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υπογραμμίζει ότι τα πιο ανεπτυγμένα κράτη-μέλη θα μπορούσαν όλο τους, το, το σύνολο των κονδυλίων τους να το χρησιμοποιήσουν εκεί που είναι ανάγκη και έτσι συνήθως τα ποσά που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη τους ή άλλως είναι πιο περιορισμένα. Επομένως, εάν ε, θέλουμε ουσιαστική απόδοση αποτελέσματος, οπωσδήποτε πρέπει να αποφεύγουμε την διάχυση των κονδυλίων σε περισσότερους στόχους πολιτικής. Γιατί να πρέπει να κατανείμουν τα χρήματα τα κρατημέλη αν ένα κράτος θέλει να επιλέξει. Από τα πιο ε, προηγμένα, ε, αν θέλει να επιλέξει παραδείγματι, να αφιερώσει όλα τα ποσά στην κοινοτομία μόνο. Και η πρόταση του εισηγητή επίσης θα επέτρεπε ε, κράτη ή περιφέρειες να ε, δαπανίσουν χρήματα στις μεταφορές, γιατί ένας από τους δύο στόχους θα ήταν οι μεταφορές, από τους οποίους θα μπορούσαν να επιλέξουν. Αλλά τα λίγα που θα μπορούν κάποια κρατημέλη να λάβουν για τις μεταφορές, για τις υποδομές μεταφορών, δεν νομίζω ότι λύνουν κανένα πρόβλημα. Ε, δύο λόγια ακόμα, αν μου επιτρέπετε, για τις παρατηρήσεις του κυρίου Φάνη Στυλρόη, διαφορά μεταξύ GNI και GDP, δηλαδή εθνικού ή εγχώριου προϊόντος. Ε, σε λίγες περιπτώσεις μόνο έχει διαφορά, λίγα είναι τα κράτη-μέλη στα οποία βλέπουμε, αλλά εμείς πάντα το GNI χρησιμοποιούμε σε εθνικό επίπεδο και το GDP σε ε, εθνικό επίπεδο. Αυτό που εννοούμε ως προς τις ε, συγκεκριμένε προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το ορίσουμε γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατανομή μεταξύ του κοινωνικού ταμείου αφενός και του περιφερειακού αφετέρου. Ε, μόνο έτσι θα μπορούμε να ξέρουμε τι χρήματα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Μια δεύτερη παρατήρηση που έχει να κάνει με τις αλλαγές που προτείνονται για τα κριτήρια αποκλεισμού Δηλαδή τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Εδώ η πρότασή μας στηρίζεται σε τρία μελήματα. Καταρχάς, ε, ότι θέλουμε συνέπεια, συνέχεια. Δηλαδή δεν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι το οποίο ήδη εφαρμόζεται. Θέλουμε συνέπεια ως προς τις νέες πολιτικές και, φυσικά πολύ σημαντικό, Οπωσδήποτε θέλουμε και να αξιοποιήσουμε την εμπειρία του παρελθόντος. Εδώ λοιπόν μας, μας απασχολούν κάποιες αλλαγές, μας ανησυχούν κάποιες αλλαγές, όπως η η πρόταση ε, για την χρήση σε τροχαίο υλικό των κονδυλίων ε, που προτείνει ο συγητής. Εμάς μας ε, κρατάει επιφυλακτικούς, δεν θέλουμε δηλαδή να ε, εμποδιστεί το άνοιγμα της αγοράς των σιδηροδρόμων, γιατί αυτό θα συνέβαινε αν εξασφαλιζόταν η δυνατότητα για χρήση των κονδυλίων αυτών εκεί. Και επιπλέον δεν θέλουμε και να περιοριστεί το πεδίο χρήσης των κονδυλίων. Και κάτι ακόμη Ε, ξέρω ότι έχετε κάπως ανάμεικτη αντίληψη ως προς τη χρηματοδότηση ορισμένων ε, πόρων σε περιοχές όπως Φερρυπίνη, Ισπανία, όπου βλέπουμε ότι δεν ε, είναι κερδοφόρα ορισμένα περιφερειακά αεροδρόμια, παραδείγματι. Ε, και έτσι δεν θα θέλαμε να δοθεί χρηματοδότηση σε αυτά και να χαθούν κονδύλια που θα μπορούσαν να πάνε αλλού ε, και πολύ πιο αποτελεσματικά. Μια τρίτη παρατήρηση που σχετίζεται με την ε, επιλογή του 5% ελάχιστη χρηματοδότηση για περιοχές με συγκεκριμένη καθυστέρηση ανάπτυξης. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα σήμαινε σημαντικό διοικητικό άχθος, ότι θα πρέπει να γίνει η διάγνωση, η σύγκριση με άλλα ε, ποσοστά και στη τελευταία ανάλυση ήταν και δύσκολο να εφαρμοσμοστεί σε ορισμένα κράτη-μέλη, δηλαδή περιοχές με συγκεκριμένο η καθυστέρηση, η ανάπτυξη στο Λουξεμβούργο, τι θα σήμαινε. Άντε και μπορώ εγώ να τις εντοπίσω, αλλά θα έπρεπε μετά να υπάρχει και μια διάταξη στη, στον κορονισμό που θα έλεγε ότι το 5% θα πρέπει να ε, δαπανηθεί για, για περιοχές συγκεκριμένη καθυστέρησης για όλα τα κράτη-μέλη και αυτό βέβαια θα άνοιγε τη συζήτηση και μεταξύ των αρχών της, υπηρεσίας, της Επιτροπής αλλά και αντίστοιχα των, κρατών, των αρχών των κρατών μελών. Δηλαδή θα έπρεπε να συνεννοηθούμε για το τι εννοούμε με τα, με τα ίδια αυτά ποσοστών. Τέταρτη παρατήρηση και συναφής με την προηγούμενη. Επίσης επιφυλακτικοί είμαστε ως προς την καταβάση, στον διπλασιασμό του ελάχιστου ποσού, ε, γιατί βέβαια αυτό ενισχύει το περίπλοκο της υπόθεσης αυτής, ε, σημαίνει επιπλέον δημοσιονομικό άχθος, και νομίζω ότι και σε αυτό το σημείο πρέπει να διατηρηθεί η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπω έχει. Επίσης, πολύ σημαντικό ε, βέβαια αλλά ίσως όχι τόσο ε, απόλυτα, ε, το επίπεδο λεπτομέρειας που έχουμε. Διότι ο στόχος μας εδώ είναι να έχουμε στόχους σύντομους, απλούς κατανοητούς, ξεκάθαρους. Άρα δεν θέλουμε να προσθέσουμε τίποτα παραπάνω σε σχέση μια, με μια ε, διάταξη που θα επέβαλε περισσότερα, περισσότερο αυστηρούς κανόνες. Γι' αυτό θα θέλαμε περισσότερη ευελιξία. Αυτό επιδιώκουμε με την πρότασή μας. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κοτσολίνο. Σε εσά η τιμή της ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης. Ας την ολοκληρώσουμε με την κατάθεση των τροπολογιών και τη δουλειά που θα κάνουμε όλοι μαζί. Εγώ επί τη ευκαιρία θέλω να πω ότι θα ήταν καλό να αποφύγουμε την παγίδα της σύγχυσης ε, των θεμάτων αυτών, δηλαδή κανονισμός εφαρμογής, ταμείο συνοχής, έτπα, να τα συστήσουμε όλοι μαζί, γιατί θα χάσουμε το στόχο μας τελικά και την εικόνα. Μια άλλη πρόταση που έχει να κάνει με το στόχο της απλούστευσης δεν πρέπει να τον συγχαίρουμε με τους πολιτικούς στόχους στην πιστοποίηση. Αν θα βάλω 6-10% δεν αλλάζει τίποτα. Απλώς έχουμε να κάνουμε μια πολιτική εκτίμηση. Ας μην μπερδεύουμε λοιπόν στόχους που προτείνει το Κοινοβούλιο, πολιτικούς στόχους, στόχους της πολιτικής λειτουργίας με την ιδέα της απλοποίησης. Μετά πολύ ευχαριστώ να συζητήσουμε τα άλλα θέματα. Η Επιτροπή θα μπορούσε να μας δώσει κάποιες βασικές ε, ιδέες έτσι ώστε να αντιληφθούμε εάν αυτό το οποίο προτείνουν ε, υπηρετεί όντως το στόχο της απλοποίησης. Και ως ε, αρκετά ειδικό στα θέματα τη περιφερειακή πολιτική και από την πρακτική μου εμπειρία, μπορώ να σα πω ότι πολλέ φορέ όταν μιλάτε εσεί για απλοποίηση, ε, μάλλον πιο περίπλοκα τα κάνετε τα πράγματα. Πολύ ευχαριστώ λοιπόν να κάτσουμε να συνομιλήσουμε, αν θέλετε, και κατηδίαν, ε, γιατί η απλοποίηση δεν ε, ε γίνεται με τα λόγια. Με τι ουσιαστικέ διαδικασίε που θα εφαρμοστούν στην κάθε περιοχή υλοποιείται η απλοποίηση. Κατά τα άλλα, πολύ ευχαριστώ. Ξέρω ότι όλοι έχουμε μέλημα την ε, πρόταση αυτή να την εμπλουτίσουμε έτσι ώστε να υπηρετήσει το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη. Και τέλει πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια καλή δουλειά, μια ουσιαστική δουλειά και με τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε και από τη συζήτηση που είδαμε βλέπουμε ότι υπάρχει γενικότερα συνένεση Περιμένω λοιπόν με χαρά τη συνεργασία με τους συναδέλφους, με την Επιτροπή. Και μέχρι το Νοέμβριο να έχουμε ολοκληρώσει εδώ στην Επιτροπή. Ελπίζω ώστε το Δεκέμβριο να μπορούμε να περάσουμε το θέμα στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν για όλα όσα συνεισφέρατε στη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Το Δεκέμβριο να ψηφίσουμε εδώ και να πάμε μετά στην Ολομέλεια. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών λοιπόν είναι 12 το μεσημέρι την 5η ε, 25 Οκτωβρίου. 22 είναι για το CPR και 25 είναι για το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ. Έτσι ευθυγραμμιζόμαστε. Καλώς. Εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη. Στα διάφορα κάτι. Παρακαλώ κυρία Κρέλ και μετά ο κύριος Φανίστεροι. Νόμιζα ότι εγώ είχα κάτι στα διάφορα, αλλά βλέπω ότι έχουν κι άλλοι. Ωραία, ακούω. Ναι, την προηγούμενη φορά στους συντονιστές αποφασίσαμε γνωμοδότηση, μάλλον όχι γνωμοδότηση για το ΣΕΦ, αλλά επιστολή. Μπορείτε να ενημερώσετε σχετικά και τη γραμματεία. Γιατί εγώ κατάλαβα ότι ετοιμάζει συμβιβασμούς, που αν πρόκειται για επιστολή δεν χρειάζεται συμβασμή. Πρόεδρος, ναι, το συζητήσαμε όντως στη συνεδρίαση των συντονιστών και θα ελέγξω τι αναφέρεται στις αποφάσεις των συντονιστών και θα φροντίσουμε. Γιατί όντως, έχετε δίκιο, συζητήσαμε τη δυνατότητα επιστολής, γιατί έτσι έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία ως Επιτροπή. Κύριε Φανίστερο, εσείς. Θα, θα έρθω μάλλον στο θέμα που θέλω να σας πω, αλλά το θυμάμαι και εγώ ότι αυτό είχαμε πει, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα με επιστολή να είμαστε έγκαιρα. Γι' αυτό, έτσι ήταν για να στείλουμε ένα μήνυμα στους προπολογισμού. Ας φροντίσουμε λοιπόν έχουμε ένα κείμενο. Για το ΣΕΦ και τη μεταφορά. Λοιπόν, τώρα εγώ δεν το ήξερα όταν ήρθα το μεσημέρι, αλλά ενημερώθηκα στο μεταξύ ότι στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας θα έχουμε και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας μας της προηγούμενης εβδομάδας, για την απόρριψη δηλαδή, στην οποία προβήκαμε των μεταρρυθμίσεων. Δεν είχα καταλάβει ότι το θέμα αυτό θα προσγειωνόταν αμέσως στην Ολομέλεια με την κυρία Μπιακόφ και υπήρχε μια άλλη πρόταση για την μπλε κάρτα που δεν συμπεριλήφθηκε γιατί οι επιτροπές δεν το δέχτηκαν και ή μπορεί το απόσυρε η μπορει το πως η επιτροπη δεν ξέρω. Μπορεί να με ενημερώσει κάποιος. Θα υπάρχει στην Ολομέλεια. Τι είδους απόφαση. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Okay. Καλώς. Όλοι είδαμε την προσωρινή ημερήσια διάταξη για την Ολομέλεια. Και το γνωρίζουμε όλοι, όλοι το είδαμε αυτό που λέτε. Η εξήγηση της γραμματείας είναι ότι είναι κάτι ουδέτερο. Η δικιά μας απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί ή να απορριφθεί από την Ολομέλεια. Υπάρχει κάτι που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη Ολομέλειας. Αν ναι, πείτε το μου να το ελέγξω. Η κυρία Κρέλ, εγώ κατάλαβα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε ένα μήνυμα απόσυρσης της πρότασης. Οπότε η ερώτηση είναι, το κάνανε? Πρόεδρος, όχι, μπορώ να ρωτήσω βέβαια την Επιτροπή. Θα μου απαντήσετε αν σας ρωτήσω. Παρακαλώ. Η Επιτροπή παρακολουθήσαμε από κοντά τις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξαρτάται από το αποτέλεσμα των δικών σας συζητήσεων. Τότε θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν και πώς θα συνεχίσει με το φάκελο αυτό παρετέρω. Προς το παρόν είμαστε σε κατάσταση αναμονής. Περιμένουμε τη δικιά σας επόμενη κίνηση όλο και βελτιώνεται, όλο και βελτιώνεται. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής μας Περιφερειακών Υποθέσεων βλέπω ότι βελτιώνεται ο συνάδελφος. Ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, προς το παρόν δεν έχουμε τίποτα παραπάνω. Άπαξ και έχω κάτι παραπάνω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα σας ενημερώσω αγαπητοί συνάδελφοι. Εντάξει, τώρα η σειρά μου. Κύριε Κρέιλ, συγχαρητήρια να σα ευχηθώ για τα γενέθλιά σα εκ μέρου ολόκληρη τη επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων. Χρόνια πολλά κυρία Κρέλ. Να ζήσετε. Έχουμε το προνόμιο να συνεργαζόμαστε με την κυρία Κρέλ, να τη γνωρίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και να συνεχίσετε να είσαστε τόσο θετικοί στις εργασίες επιτροπής μας. Τίποτα άλλο δεν είχα για τα διάφορα μόνο. Να υπενθυμίσω, επόμενη συνεδρίαση που θα είναι πάλι έκτακτη θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο την 5η 25 Οκτωβρίου. 10 και 4. 10 και 4. τη ρώτησε η κυρία Κρέλ χωρίς μικρόφωνο, απάντηση, θα το προσπαθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος. Λύεται η συνεδρίαση.